start Καλημέρα σας. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε, διότι έχουμε μόνο μία μισή ημέρα συνεδρίασης. Καλωσορίζω όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ως προς το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, όπως ε, σας έχουμε ήδη ενημερώσει, Αλλάξαμε σειρά σε κάποιες εκθέσεις. Έχουμε την κυρία Κανιέτη για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή και την κυρία Λεγκρίπ για τον ενωσιακό τελωνιακό κώδικα. Θέλανε να αλλάξουν τη σειρά και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, οπότε θα αρχίσουμε με την κυρία Κανιέτη. Ένα λεπτάκι θα επανέλθω σε αυτό. Σήμερα το απόγευμα έχουμε πάρα πολύ σημαντική ακρόαση σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η κυρία Βερνιό θα είναι συντονίστρια. Ελπίζω να υπάρξει αθρώα προσέλευση. Εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ωραία. Κάποιες ανακοινώσεις πρωτού ξεκινήσουμε. είχα την τιμή να λάβω μία πρόσκληση από τη διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, των Εθνικών Κοινοβουλίων εννοώ, την ΚΟΖΑΚ δηλαδή, ε, την Κυριακή και τη Δευτέρα ήμασταν στην Κοπενχάγη και παρουσιάσαμε τις εργασίες μας για την εσωτερική αγορά. Έτυχε θετικότητα της υποδοχής, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, ε, τόνισα πόσο εκτιμούμε τη συμβολή των Εθνικών Κοινοβουλίων στις εργασίες μας και θα εντείνουμε την συνεργασία. Ε, και ήμασταν στο ίδιο πάνω με τον κύριο Μπαρνιέ και ακούσαμε τις ερωτήσεις μαζί. Άλλαξε λίγο το σενάριο, γιατί συνήθω εγώ είμαι πρόεδρος, είναι δίπλα μου ο κύριος Μπαρνιέ και όλες οι ερωτήσεις απευθύνονται προς αυτόν. Τώρα έλαβα και εγώ ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και προβάλαμε και το έργο της Επιτροπής μας. Χαρήκαμε που αναγνωρίστηκε δεόντω ε, η συμβολή μα από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα εκπονήσουμε και έκθεση των πραγμένων και οποιοδήποτε έγγραφο προκύψει θα σας το διαβιβάσουμε. Η γραμματεία της ΚΟΖΕΚ ε, εκπώνησε δύο συνόψεις ε, για τα πραγμένα στην εσωτερική αγορά για τα, τους 12 μοκλούς της εσωτερικής αγοράς και ο κύριος Μπαρνιέ μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται μια νέα δέσμη προτάσεων για να ενισχύσει την πράξη για την ενιαία αγορά μέχρι το 2013. Ελπίζω σήμερα το απόγευμα οι συντονιστέ να το συζητήσουν αυτό το θέμα για να τοποθετηθεί και η Επιτροπή μα εν ώψη τη διαδικασία. Αυτά για τη συνεδρίαση τη ΚΟΖΑΚ. Δεύτερον, χαίρομαι ε, που σας ανακοινώνω ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας όπως και όλες. Και έχουμε ένα νέο newsletter, ενημερωτικό σημείωμα της ΙΜΚΟ, έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Ε, έχετε και τους διαδικτυακούς συνδέσμους όταν το επισκέφτεστε επιγραμμικά και μπορείτε να έχετε όλη την τεκμηρίωση, οπότε θα το δείτε στην ιστοσελίδα και θα παρακολουθεί οποιοδήποτε, όχι μόνο τα μέλη της Επιτροπής, τις εργασίες ε, της ΙΜΚΟ. Επίσης, να υψίσετε την προσοχή σα στο ότι μέσα στους φακέλους η γραμματεία μας που εργάζεται τόσο σκληρά μας προετοίμασε τα περί της νομολογίας ε, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις εκχωρήσεις μάλλον για τις παραχωρήσεις. Ε, είχαμε και ένα σχετικό εργαστήριο για τις παραχωρήσεις. Το έχουμε προγραμματίσει για τις 10 Μαΐου το απόγευμα, έτσι δεν είναι. Ούτως ή άλλως θα σας στείλουμε υπενθύμηση. Θα συζητηθούν κάποια ζητήματα, ο κύριος Ζήμαν θα συντονίζει για να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με θέσει τη Επιτροπή μα, πώ δηλαδή θα αντιδράσουμε στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι παραχωρήσει. Αυτά λοιπόν για τι ανακοινώσει και σχέση με τα πρακτικά. Θα πω μόνο ότι έχετε μέσα στου φακέλου σα πρακτικά για, τις, για δύο συνεδριάσει τον Οκτώβριο πέρσι και μία από το Μάρτιο φέτο. Θα έχετε διαβάσει υποθέτω τα πρακτικά. Αν δεν προβάλλετε ένσταση μέχρι το πέρα συνεδρία, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Ε, περνούμε τώρα στο πρώτο σημείο. Ε, είναι η έκθεση της κυρίας Καλνιέτη, η γνωμοδότηση μάλλον της κυρίας Καλνιέτη για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές σημείο 16. Ο Άντερς Φάμπερς ε, θα αντικαταστήσει την κυρία Καλνιέτε. Ο κύριος Σίβιτς είναι ο Σκιώδης. Εδώ είστε, καλωσορίσατε κι εσείς. Από τους σοσιαλιστές η κυρία Ρούλε, ε, πράσινη. Ο κύριο Κλωσινέσκι θα μιλήσει από πλευράς του κυρίου Μπίλνε. Ναι. Θα τα βρούμε μεταξύ μας. Με τα χαράς. Καλωσορίζω τον κύριο Βενουά ε, που ε, είναι στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς στο Τμήμα Ενέργειας θα σας ακούσουμε μετά τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητέ. Κύριε Σβάντο, παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κάιμη η οποία για προσωπικούς λόγους δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα και όσον αφορά την εισαγωγή της θα την παρουσιάσω εγώ για λογαριασμό της και ε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη διότι η συνεργασία για την για ε, ε, την προώθηση ήταν ε, πολύ πολύ καλή. Βεβαίως υπήρξαν διάφορες τροπολογίες τις οποίες θα προσπαθήσει να ενσωματώσει αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει για όλες διότι θα περιοριστεί ιδίω στη δικιά μας δικαιοδοσία και σαν εκπρόσωπος των Πρασίνων θα ήθελε να τονιστεί η περιβαλλοντολογική πτυχή και επίσης η κυρία Καλνιέτε που έχει και μία άλλη γνωμοδότηση ε, θα ήθελε ουσιαστικά να περιλάβουμε και θέματα που είναι σημαντικά ε, για την, αγορά, για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών. Αλλά θα ήθελε να έχουμε μία πλήρη ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη το ταχύτερων δυνατόν χωρίς ε, μέσα στο δίκτυο αυτό να αισθάνεται μία χώρα απομονωμένη στην ενιαία ενεργειακή αγορά διότι εδώ είπαμε ότι θα χρειαστούν 200 δισεκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθεί το δίκτυο αυτό κατά τρόπον όλοι, ώστε όλοι οι πολίτες όλων των κρατών μελών να είναι εξασφαλισμένοι ότι θα έχουν ενεργειακή ασφάλεια η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να έρθει ιδίω από τον ε, ιδιωτικό τομέα. Επιτρέπεται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι από τις τρίτες χώρες και η κυρία Καλνιέτε μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί διότι βεβαίως υπάρχουν διάφορα νομοθετικά μέτρα που πρέπει να συνυπολογιστούν όπως παραδείγματος χάρη το νομικό μέτρο ε, για την συμφωνία για τις δημόσιες αγορές ε, ε, τα μέτρα αυτά προβλέπονται και έχουν δεσμευτεί 9 δισεκατομμύρια για το στόχο μας στην επόμενη δημοσιονομική ε, πρόβλεψη και βεβαίως ε, ε, τα 9 μέχρι τα 200 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και αντιλαμβάνεστε ότι αν πρόκειται για μικρά προγράμματα δεν θα ενδιαφερθούν οι ιδιώτες. Αλλά η κυρία Καλνιέτε ιδίω επικεντρώνεται ή στην συμμετοχή των καταναλωτών και αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για αυτήν και αυτό το είπε σαφώς και στην γνωμοδότηση ήταν ότι ε, οι καταναλωτές στις απομακρυσμένες περιοχές θα χρειαστεί να καταβάλουν υψηλότερες τιμές για την ενέργεια ε, και θα έπρεπε κατά τη γνώμη της να εξασφαλίσουμε να μην αυξηθούν οι τιμές της ενεργείας διότι ουσιαστικά είναι ένα ε, βασικό στοιχείο στοιχείο του κόστους διαβίωσης και πρέπει να προσπαθήσουμε η ε, τροφοδότηση με ενέργεια να είναι εφικτή για όλους τους καταναλωτές Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά είχα να πω σήμερα για την ε, γνωμοδότηση της συναδέλφου κυρίας Καλνιέτε. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 7 Μαΐου και η καθηγήτρια σας ε, καλεί να διατυπώσετε προτάσεις ή τροπολογίες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ ότι η κυρία Καλνιέτε έχει δίκιο διότι εντοπίζει όπως είπατε σε την γνωμοδότησή της σε θέματα που μας ενδιαφέρουν ε, για την Επιτροπή αυτή παρόλο που υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο για την πρότασή της που και αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Σίβιτς τώρα θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ε, ευχηθώ καλή ανάρρωση στην εισηγήτρια διότι η έκθεση δεν ε, την εμπόδισε ίσως να έρθει αλλά, τώρα αλλά έχει συγκεντρώσει τις απόψεις ολονών μας και κατόπιν αυτού έχουμε μία έκθεση η οποία δεν είναι πολύ αντιφατική πράγμα που είναι σπάνιο εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος θα ήθελα να αναφερθώ σε την ιδιομορφία αυτού του θέματος γιατί είναι εύκολο να ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και θέλω εδώ να επισημάνω τρία θέματα που μας απασχολούν στην ανάλυση μας. Καταρχήν ότι είναι σαφές βήμα προς την ενιαία αγορά. Για πολύ καιρό ε, είχαμε πει ότι η ενιαία αγορά είναι ένα απόμακρο όνειρο ε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και αν, ε, αν δεν υπάρξει υποδοχή υποδομή δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία αγορά. Είναι δηλαδή ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πρέπει όμως να σας πω ότι υπάρχουν τρεις ενεργειακές πηγές. Ε, ε, ε, το πετρέλαιο, το αέριο και όλες οι άλλες μορφές. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους τελικούς καταναλωτές και αποδέκτες, διότι μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια και εδώ εξετάσαμε το θέμα της ασφαλείας των τελικών καταναλωτών από άλλη οπτική γωνία, διότι ο κύριος Βόμπα αναφέρθηκε στο θέμα της τιμής, ενώ εμείς θέλουμε να πούμε ότι άπαξ και καταρτιστεί αυτή η υποδομή, οι τιμές ενεργείας θα έπρεπε να μειωθούν. Δηλαδή δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα μέλη της Επιτροπής μας να επιτευχθεί. Επίσης, το θέμα της τιμής είναι κάτι που μας ε, ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και από αυτή την οπτική γωνία η αύξηση και βελτίωση του δικτύου ενεργείας είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πακέτο το οποίο ε, βλέπουμε εις τις τροπολογίες ε, του εισηγητή θα μπορέσει να διευρυνθεί με επιπρόσθετα στοιχεία στην οποία περίπτωση θα το συζητήσουμε με την κυρία Καρνιέτε. Θέλω όμως εδώ να αναφερθώ και σε κάτι άλλο ακόμη. Ε, δέχεται να μην προέκυψε στη δικιά μας επιτροπή αλλά έχει προκύψει στα εθνικά κοινοβούλια. Το θέμα της ε, γραμμής των πιστώσεων που λέγεται έχει επικεφαλίδα Connecting Euro μπορεί να αποτελεί μία απειλή για την πολιτική συνοχής. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ακόμη και αν δεν είναι στη δικαιοδοσία της δικιάς μας Επιτροπής δεν θα πρέπει αυτά να συμβούν βάρος της πολιτικής συνοχής γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο ιδίως αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ εύστοχα τα σχόλιά σας. Θα δώσω το λόγο και στην Επιτροπή να μας πει λίγα λόγια για το πώς συνδέεται αυτό με την πολιτική συνοχή όπως είπατε, κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η κυρία Καλνιέτε ευτυχώς ε, έχει περιοριστεί στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας ε, σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα διότι δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να ασχοληθούμε με την χρηματοδότηση των δικτύων πράγμα που είναι αρμοδιότης άλλων επιτροπών. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις αρμοδιότητες της δικιάς μας Επιτροπής, γι' αυτό και συμφωνώ με τα σχόλια από τις πλευράς περιβάλλοντος αυτό που προσπαθούμε είναι να μην αντιταχθούμε και να μην μπούμε στα μπελοχώραφα των άλλων επιτροπών, πράγμα το οποίο έκανε η κοινία Καρνιέτε και συμφωνώ απολύτω με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος παρακαλώ, κάποιος άλλος συνάδελφος να τοποθετηθεί. Ο κύριος Σίβιτς, θέλετε να το πω και πάλι. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα μεταφραστικό και δεν πέρασε καλά το μήνυμα με εγώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το θέμα. Και απλά μετέφερα ένα μήνυμα που έμαθα μια είδηση από τα Εθνικά Κοινοβούλια που πιστεύω ότι είναι προς όφελος όλων να το γνωρίζουν, ότι είμαι ε, κατά της διεύθυνσης αυτής. Ελπίζω να πέρασε το μήνυμά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βενουά, θέλετε να κάνετε τα σχόλιά σας. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Σουάπ που αναπλήρωσε την κυρία Καλνιέτε στην παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Η έκθεση αυτή πραγματικά εστιάζει στι αρμοδιότητες της Επιτροπής σας και θα έλεγα ότι όταν μιλάμε για ενεργειακέ υποδομές είμαστε ακριβώς στον τομέα αρμοδιότητά σας. Γιατί χωρές ε, υποδομές δεν έχουμε ιστορική αγορά. Αυτή είναι η ουσία σήμερα. Και βλέπουμε πραγματικά ένα έλλειμμα υποδομών που δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε στην ολοκλήρωση των 27 ενεργειακών αγορών σε μια ενιαία ενεργειακή αγορά, από την οποία θα έχουν πολλά ωφέλη οι καταναλωτές. Το πρώτο όφελος θα είναι οι πιο ανταγωνιστικές τιμές, πράγματι. Όταν βλέπετε τις διαφορές των τιμών, κατά 30% ανάμεσα στις χώρες ανατολική Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης, αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, είναι απαράδεκτο σε μια ενιαία αγορά. Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη υποδομών. ιδίω, γιατί υπάρχει ένας κυρίαρχο πάροχος σε αυτές τις χώρες, κάποιες φορές είναι και ο μόνος πάροχος σε αυτές τις χώρες που υποδεικνύει τις τιμές, και αυτή η κυρίαρχη θέση, δεσπόζουσα θέση που υπάρχει πολύ συχνά, δεν μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανταγωνιστικές ε, τιμές. Οι υποδομές αυτή τη στιγμή αποτελούν μόλις το 5 έως 10% της τελικής τιμής που φτάνει στο καταναλωτή. Άρα λοιπόν η απροθυμία για την κατασκευή νέων υποδομών όπου αυτό είναι αναγκαίο και επιμένω όπου είναι αναγκαίο γιατί λέμε ότι χρειάζεται μία εύρωστη μελέτη α, κόστους οφέλους για να προβούμε σε νέες κατασκευές. Τότε οι επενδύσεις υποδομές θα επηρεάσουν πάρα πολύ την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί με αυτό το 5-10% που σημαίνει υποδομή στην τελική τιμή, αυτό μπορεί να επηρεάσει κατά 40-50% την τελική τιμή ε, του βασικού αγαθού που πληρώνει ο καταναλωτής. Οπότε μιλάμε για μια πολύ σημαντική επένδυση. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε και είναι πολύ σημαντικό είναι η έλλειψη κατανόηση σχετικά με την ανάγκη για τον ίδιο υποδομέ. Πολλοί λένε όχι εδώ δίπλα μου, όχι σε μένα εδώ στην πόλη μου, στη γειτονιά μου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα γενικότερη αποδοχή αυτών των υποδομών. Και τέλο πρέπει ο καταναλωτή να αποφασίσει. Θέλει ασφάλεια στην παροχή ενέργεια. Αν το θέλει, χρειάζονται υποδομές. Είναι κάτι λοιπόν πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν όλοι. Γιατί είναι το θέμα, εν προκειμένου, είναι ο τρόπος λειτουργίας του ενεργειακού συστήματο και ιδίω ε, ε, του εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό. Και στο μέλλον αυτό θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο. Αν δεν έχουμε τι κατάλληλε υποδομέ, θα υπάρχει ο κίνδυνο της διακοπής, των διακοπών γενικότερα ε, της παροχή. Και αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές. Θα πρέπει, αν θέλετε, να ενημερώσουμε το καταναλωτή. Αυτό είναι κομμάτι ε, καθαρά της πολιτικής εσωτερικής αγοράς και κατανοώ την ανησυχία της κυρίας Καλνίτ όπως εκφράζεται στην έκθεση. Ποια είναι τα ωφέλη για τον απλό καταναλωτή. Με άλλα λόγια, ο σωστός όρος θα ήταν το νοικοκυριό. Τα νοικοκυριά είναι εν προκειμένου αυτό, αυτή η ομάδα στόχος. Μα τα νοικοκυριά είναι, αν θέλετε, οι δικαιούχοι αυτοί που υποφελούνται από όλες αυτές τις πολιτικές και τη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε λοιπόν ότι εργαζόμεθα προς την επίτευξη των στόχων που όρισαν οι ενεργοί κρατών κυβερνήσεων. Πέρυσι, το Φλεβάρι του 2011, υπήρξε η απόφαση να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αγορά στο 2014. Και να ε, υπάρξει και η σχετική διασύνδεση και των ε, νήσων στην ενιαία αγορά μέσα στο 2014. Όλα λοιπόν που συζητούμε σήμερα θα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, το SAFE. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει καμία επικάλυψη με την πολιτική συνοχής και ε, το Ταμείο Συνοχής, το ΣΕΦ, το CEF, καλύπτει τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, οπότε είναι στο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας αυτό το ταμείο. Η πιθανή λοιπόν επικάλυψη με τα περιφερειακά ταμεία, ναι, είναι κάτι που να συζητήσουμε, αλλά όχι με τη συνοχή. Τώρα, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πραγματικά, μια γνήσια ευρωπαϊκή προσέγγιση υποδομές. Γιατί μπορεί να χρειάζεται να κατασκευαστούν υποδομές σε μια χώρα που να ωφελήσουν τελικά τη γειτονική της χώρα. Αν ρωτήσετε τώρα τους TSO αν θα το κάνουν αυτό, θα σου πούνε όχι. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα ε, συνολικό και ρυθμιστικές αρχές που ορίζουν τα τιμολόγια να κάνουν μια σωστή κατανομή του κόστους και τους ωφέλους αλλά αυτό κάποιες φορές δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν ε, υποδομές εολικής ε, υπεράκτιας ενέργειας και βλέπουμε ότι αυτές οι υποδομές είναι κατά κύριο λόγο στην, ε, στη Βόρεια Ευρώπη. Όμως αυτή η ενέργεια που γεννάται είναι προς όφελος όλες τη Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης. Χρειάζεται λοιπόν κίνητρα. Αν μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε αυτά τα project θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια ευρώ και θα εξοικονομήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Αυτό είναι λογικό γιατί είναι κάτι που θα είναι προς όφελος όλων και των καταναλωτών. Άρα χρειαστεί λοιπόν να έχουμε έναν κουμπαρά αν θέλετε, όπου να βάζουμε χρήματα για να χρηματοδοτούμε τα εκφύσεως αν θέλετε, διαμεθοριακά προγράμματα που κάποιες φορές α, ωφελούν πιο πολύ μια χώρα και όχι το στην άλλη. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποια χώρα ε, ωφελεί περισσότερο ένα πρόγραμμα. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα που να ωφελεί κάποιον 40%, έναν άλλον 20% και έναν 5%. Όμως αν θέλουμε ολοκλήρωση αγοράς και θέλουμε εξασφάλιση του εφοδιασμού ε, του καταναλωτή, μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι καθαρά ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν είναι καθόλου εθνική προσέγγιση. Γι' αυτό υπάρχει σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με το πώ χρησιμοποιούμε το Περιφερειακό Ταμείο. Αυτά ευχαριστώ. Well, thank you. Thank you very much, uh, for... Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμη η επισκόπηση του προγράμματος και μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε μία από τις αρμόδιες επιτροπές. Έχουμε λίγο χρόνο. Δεν θα έρθει η κυρία νομίζω μέχρι τις 10. Ο κύριος Μάντες όμως είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κι εσείς κάτι γιατί ο σκιώδης σας δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μάιερ ναι, είναι γεγραμμένος ήδη στον κατάλογο μας. Ε, θα κάνουμε άλλον ένα γύρο παρεμβάσεων μετά και την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Σφάμπ, η κυρία Φερχάινες από την Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξης είναι εδώ, σας καλωσορίζω. Ξέρω ότι ειδικεύεστε στα θέματα, τα περιφερειακά θέματα. Κύριος Μαΐ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να αφαιρθώ σε δύο θέματα εν συντομία. Καταρχήν την κατάρτιση των δικτύων, τα οποία ιδίω για τις ανανεώσιμες ενέργειες πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά από ό,τι τα ισχύοντα. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται εις τις εγκαταστάσεις στην Βόρειο Θάλασσα, η οποία δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα, τα, τα στοιχεία που βρίσκονται στην ξηρά και υπάρχει πρόβλημα αν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την ενέργεια που παράγεται και αυτό δεν πλήττει μόνο την κάτω Σαξονία και τη Γερμανία αλλά και γειτονικέ χώρες. Δεύτερον, όσον αφορά τις τιμές, όταν υπάρχει μια διαφορά τιμής 30% δεν οφείλεται στην υποδομή σε έλλειψη δικτύων αλλά οφείλεται σε πολιτικούς παράγοντας διότι στη Γερμανία ε, το ίμιση της τιμής ενεργείας ε, είναι η τιμή της ενέργειας και το άλλο μισό τίμημα της πολιτικής και αυτό επηρεάζει τις, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας δεν έχει να κάνει δεν έχει σχέση με τα δίκτυα αλλά και δεν πρόκειται να βοηθήσει στην επέκταση της υποδομής των ανανεωσίμων πυρών ενεργείας. Πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχήν τι κοστίζει και πώς μπορούμε να καλύψουμε το κόστος και δεύτερον να έχουμε υπόψη μας ότι οι ενεργειακές τιμές ε, διαμορφώνονται ακόμη βάσει ε, εθνικών κριτηρίων και όχι βάσει των κριτηρίων της εσωτερικής αγοράς. Η κυρία Ρούλε ε, θέλει πάλι το λόγο. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Μάγερ είπε τα περισσότερα που ήθελα και εγώ να πω, αλλά θέλω να τονίσω ένα θέμα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Είμαστε υπέρ, πλήρως υπέρ ε, της ε, ε, στηρίξεως των ευρωπαϊκών δικτύων και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε απλώς διεθνικά δίκτυα αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε μετακομίσουμε τις ε, αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής από τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ήτρε ή κάποιας άλλης Επιτροπής. Ο κύριος Σίβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σχολιάσω την παρουσία του εκπρόσωπου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας μίλησε για την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του προγράμματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταρρεύσουν ε, κάποια στερεότυπα, να καταρρύψουν μάλλον κάποια στερεότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικρατεί η άποψη ότι αν περιορίσουμε τη δράση των διαρθρωτικών ταμείων, αυτό σημαίνει ότι θα καταργηθούν και τα σχετικά κονδύλια. Με τη θετική σας όμως επιχειρηματολογία βλέπουμε κάτι πολύ λογικό ε, να διαγράφεται. Φυσικά δεν γίνεται να προχωρήσουν τέτοια προγράμματα σε μεμονωμένη βάση. Υπάρχουν ε, πολλές ε, πολλά εθνικά προγράμματα, αλλά η ολοκλήρωση δεν μπορεί παρά να πραγματοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. για το 2014 ως 20 ε, την επόμενη περίοδο θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει, να μην περιμένει. Ε, συνεχίστε με αυτή την θετική σας άποψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σφάπ ε, θέλει να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Κύριος Μάντελς πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη γιατί κόλλησα στην κίνηση, αλλά συμβαίνουν αυτά. Όλες την ο Σκιώδη εισηγητή ε, και μου είπε να παρέμβω τουλάχιστον για κάποια ζητήματα και να θέσω ερώτηση προ τον εισηγητή. Πρόκειται για μια προσθήκη. Ordinary consumers, αυτή η έννοια του συνήθους καταναλωτή. Τι σημαίνει αυτό, θα μπορούσε να επεκταθεί ο εισηγητή. Ε, λέει όλε τι αυροφροσύνε, δεν χρειάζεται να τα πω και εγώ, τα ακούσαμε από του άλλου, θα περάσω στην ουσία. Κάποιες τροπολογίες θέλουμε να προσθέσουμε για να ενισχύσουμε την περαιτέρω τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αποφύγουμε την στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Αυτά ήθελε να πει ο κύριος Όλε Σμιτ και εγώ θέλω να προσθέσω κάτι σε σχέση με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σε κάποια άρθρα βλέπω ότι η τιμή της οικοδόμησης νέας υποδομής σε κάποια μέρη της Ευρώπης κοστίζει πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Άρα, για να αποφασίσουμε, θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το επιπρόσθετο κόστος, ε, δηλαδή είναι πιο περίπλοκο. Ε, ένας αυτοκινητόδρομος στην Ελβετία μπορεί να κοστίζει πολύ περισσότερο από έναν αυτοκινητόδρομο στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και πάντοτε προσπαθώ να βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι. Για να είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν και να παραμείνουμε αισιόδοξοι θα πρέπει να διερευνήσουμε, να δούμε ε, πώς αιτιολογούνται αυτές οι επιπρόσθετες επενδύσεις, κυρίως επειδή πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Για την ενέργεια πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καθολική πρόσβαση για όλους. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Σουβάμπ. Ε, ήθελε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, να δευτερολογήσει. Έχουμε χρόνο, άμα θέλετε να απαντήσετε τώρα στι ε, παρατηρήσει στο μέλλον τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολύ καλό που έχουμε χρόνο εδώ στην Επιτροπή για να εξηγήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Για τα δύο-τρία ερωτήματα που μου έθεσαν στον δεύτερο γύρο, θα έλεγα το εξή. Για το κόστος οικοδόμησης και τα μέτρα σύγκρισης, φυσικά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και οι νομοθετικές αρχές είναι εθνικές ε, και πρέπει να εγκρίνουν τις επενδύσεις ε, που προτείνουν οι προμότες, οι κατασκευαστικές εταιρείες. τώρα έχουμε και την υπηρεσία για την συνεργασία των εθνικών ενεργειακών ε, αρχών. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σώμα και νομίζω ότι μπορεί να γίνουν οι έρευνες κάλλιστα και να δούμε γιατί υπάρχει διαφορά στο κόστος. Όντως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Για τις ανανεώσιμες Έχουμε εθνικά ε, συστήματα υποστήριξης και τον Ιούνιο, θα, αν δεν κάνω λάθο, θα εκδώσουμε ανακοίνωση για τα προγράμματα στήριξης για τις ανανεώσιμες και θα μεριμνήσουμε ώστε τα συστήματα, τα καθεστώτα αυτά θα συγκλίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού. Φυσικά στην εσωτερική αγορά ενέργεια. είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρη κατανόηση ε, του τι ισχύει τη σημερινή μέρα για τις ανανεώσιμες, τι μπορούμε να κάνουμε και όσο περισσότερες ανανεώσιμες ε, έχουμε στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τόσο πιο ευέλικτα και πιο, διασυνδεδε... πιο ευέλικτες και πιο διασυνδεδεμένες υποδομές ε, θα χρειαζόμαστε. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο διακύβευμα. πρέπει να βέλτιστοποιήσουμε τις ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Αυτό σημαίνει ότι όπου έχουμε τον αέρα να έχουμε την αιωλική, εκεί όπου έχουμε τον ήλιο να έχουμε την ηλιακή και να αποφύγουμε ε, την χρηματοδότηση ανανεώσιμων εκεί που δεν φυσάει ο αέρας και δεν έχουμε και πολύ ήλιο. Είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους ε, και νομίζω ότι από ευρωπαϊκή απτική γωνία θα πρέπει να κάνουμε τα δέοντα για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των ανανεώσιμων. Θα σταματήσω εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ε, τις ε, σκέψεις που μας κοινοποιήσατε που τροφοδοτούν και το δικό μας προβληματισμό. Ευχαριστώ κύριο σε Μία επερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για πόσο καιρό θα χρειαζόμαστε ακόμη τα ορυκτά καύσιμα Περνάμε τώρα στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τι κάνουμε, επενδύουμε για την υποδομή και σε 20-25 χρόνια δεν χρειαζόμαστε καν ε, ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα. μπω πάνε στράφει όλε αυτέ οι επενδύσει. Yes, thank you very much. Um, well... Ναι, να σα απαντήσω. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι μια καλή πολιτική είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση. Αν είδατε το νοδικό χάρτη για την ενέργεια στο 2050 Εκεί εξετάζουμε πολλά σανάρια για το πώς δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί το ενεργειακό σύστημα την επόμενη 40 ετία. Βλέπουμε ε, μεγαλύτερη ηλεκτροποίηση, αν θέλετε, του ενεργειακού συστήματο. Κατά κύριο λόγο, η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. όμως ο άνεμος και ο ήλιος δεν είναι πάντοτε παρόντες, οπότε πρέπει να συνδυάζουμε αυτές τις πηγές με άλλες πηγές. Εκεί λοιπόν το φυσικό αέριο δίνει τη μεγαλύτερη ε, δυνατή ευελιξία ώστε να υπάρχει ένα συνδυασμός με τις ανανεώσιμες. Στον ειδικό χάρτη λοιπόν για το 2050 θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ιδίως το φυσικό αέριο τις επόμενες δεκαετίες και όσοι αφορά τα ορυκτά καύσιμα ναι, θα υπάρχει μια ανάγκη για να απομακρυνθούμε όλο και περισσότερο από τον άνθρακα έως το 2030. Ξέρετε, ήμασταν πολύ αισιόδοξοι. Πριν από πέντε χρόνια μιλάγαμε για το 2020. Όμω ε, η τεχνολογία δέσμευση και αποδίκευση του άνθρακα τελικά ε, δεν έχει δώσει πλήρω τα αποτελέσματα ακόμη. Οπότε χρειάζεται να απελευθερωθούν από τον άνθρακα ε, τα ορυκτά καύσιμα, αν θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε στον διακόμιγμα του μέλλοντο. Όμως, δεν μπορούμε πολύ απλά να καταργήσουμε μια ενεργειακή πηγή έτσι απλά. Πρέπει μάλλον να χρησιμοποιούμε όλες τις πηγές που έχουμε, αρκεί να μπορούμε να έχουμε μια δυναμική μετάβαση σε μια ε, ενέργεια με χαμηλή χρήση άνθρακα. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που ήσασταν παρόν στη Συνήθεια τη Επιτροπή μα. Ήταν εξαιρετική ευκαιρία. Ε, δεν είναι συχνό φαινόμενο κάποιο ανώτερα ιστάμενο από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ενέργεια να είναι σε εργασίε μα. Ο κύριο Φαπ θα ήθελε να κλείσει συνοπτικά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσον αφορά του βασικού στόχου έχουμε συμφωνήσει ε, διακομματικά και ε, ο στόχος μας είναι να υπάρχει ενιαία τιμολόγηση διευρωπαϊκά και να πιέσουμε τα trust της ενεργείας προς αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν απευθύνεται μόνο στα νέα κράτη-μέλη αλλά και ε, τα παλιά κράτη-μέλη μεταξύ του ΚΕΛ και του Στρασβούργου δίπλουν, λείπουν ορισμένες συνδέσεις οι οποίες οφείλονται στα μονοπόλια της ενεργείας και αυτή είναι μια σημαντική ανησυχία μας. Αν το συμφωνήσουμε είναι κάτι που θα με ικανοποιήσει. Νομίζω ότι η κυρία Κανιέτε βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι αυτά τα οποία είπα για τους καταναλωτές, για τους πολίτες ή όπως μας διόρθωσε η Επιτροπή για τα νοικοκυριά τα οποία καταναλώνουν την ενέργεια θα μας επιτρέψουν να έχουμε μέχρι τις 7 Μαΐου τις τροπολογίες για να μπορέσει να προωθηθεί η έκθεση στην Ολομέλεια για ψηφοφορία. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται και από τη συζήτηση πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το ζήτημα. Η κυρία Καλνιέτε και η γνωμοδότησή τη, νομίζω ότι θα το αντικατοτουρήσει αυτό το ενδιαφέρον. Αυτό που ο κύριος Βεβ για την ανάγκη απόδοσης κινήτρων ώστε να οικοδομηθούν αυτές ε, οι διευρωπαϊκέ Ελληνικέ υποδομέ ώστε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα η εσωτερική αγορά προ όφελο του καταναλωτή, αλλά και γιατί η παραγωγή α, ανώσιμων πηγών ενέργειας ε, ποικίλει από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή και αυτό ιδίω αφορά την Νότια Ευρώπη που ε, είναι πιο οξύς και κατά καλοκαίρια και ε, η εποχική ζήτηση ποικίλει σημαντικά. Σας ευχαριστώ πολύ τη Σάντρα, παρότι να πούσα και ευχαριστώ βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρουσία της. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή είμαστε αρκετά μπροστά ε, στο χρόνο, γιατί ήσασταν εσείς πολύ συνεπείς, να πω ότι περιμένουμε ακόμη τον ε, κύριο Αρία Σετσεβαρία, που είναι το επόμενο σημείο στη διατάξη, οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή έως τις 10, να πιούμε ένα καφεδάκι ή να τα πούμε με τους συναδέλφους μας. Και όταν ο κύριος Αρίας είναι εδώ, στις 10 ακριβώς, θα ξεκινήσουμε αμέσως με, το, με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Uh, so, ladies and gentlemen, we are ready to resume. Our rapporteur is here. Κυρίες και κύριοι, να ξαναρχίσουμε καθώς ο κύριος Αρίας έχει φτάσει. Good. So, come... Λοιπόν, να καλωσορίσω τους συναδέλφους που τώρα ε, προσήλθαν σε εργασίες της Επιτροπής μας για τη συζήτηση ενό πολύ σημαντικού σημείου. Είναι μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, μάλλον μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, σε απάντηση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση ενιαίας ψηφικής αγοράς. Ξέρετε ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς έχει τοπιστεί ως κύρια προτεραιότητα στα προγράμματα ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Και όπως είπα και νωρίτερα, ε, πραγματικά αισθανόμαι προνόμιο μου να ε, έχω λάβει αυτή την πρόσκληση για να συμμετάσχω και να είμαι ομιλητή στη διάσκεψη των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπενχάγη την επόμενη Δευτέρα. είναι ένα θέμα που μου απασχολεί όχι μόνο εμένα και πολλούς συναδέλφους. Τώρα να ευχαριστώ τον Παύλο Αρίες και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για αυτή την έκθεση. Η ομάδα εργασίας συνεδρίασε αρκετές προς το τελευταίο τρίμηνο. Ε, υπήρξε αθρώα προσέλευση συναδέλφων όπου έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσει. Η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποια όρια μέγιστης, μέγιστου αριθμού σελίδων κτλ υπάρχουν και οι σκιώδες που θα έχουν να πούν λίγα λόγια. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλία ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο και ζητά τροποντινά την πρόταση, την επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ψυχικής αγοράς. Επίσης, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές όπως είναι η ατζέντα του καταναλωτή, που από ό,τι ξέρουμε στις 22 Μαΐου περιμένουμε τη σχετική ανακοίνωση από την Κομισιόν και θα περιέχει σημαντικά στοιχεία που αφορούν το ρόλο του καταναλωτή στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Πολλά πράγματα λοιπόν αναμονή και έπειτα η έκθεση της κυρίας Πίτ για την ελληνική πώληση εμπεριέχει πολλά στοιχεία για το θέμα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Και να πω ότι στο τελευταίο workshop για την ενιαία ψηφιακή αγορά είχαμε πολλούς εκπροσώπους από βρετανικές κοινοπραξίες και από άλλους ε, παρόχους ε, ε, που παρέχουν τις υπηρεσίες επιγραμμικά. Θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται στο πολύ συχνά. Είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και καλό τον εισηγητή τον κύριο Αρίας να ξεκινήσει τη συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Μάλκομ. Θα ήθελα να έχω φτάσει νωρίτερα συνεδρίαση, όμως δυστυχώς είχα μια άλλη συνεδρίαση και δεν μπορούσα να την κλείσω εγκαίρως. Προσπάθησα να είμαι στην ώρα μου πάντως ε, και λυπάμαι που σας καθυστέρησα λιγάκι και αναγκαστήκατε να διακόψετε τη συνεδρίαση. Θέλω να ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι χειροκροτούμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία, όπως γνωρίζετε, συνεργαζόμαστε στενά επί του θέματος. Είναι μια πρόταση αυτή που, αν και η... πολύ καλή, αν και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Υπάρχει ένα δυναμικό 500 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πούμε ότι οι συναλλαγές μέσω ίντερνετ δεν λειτουργούν σε με πλήρε δυναμικό. Και ενώ στην Ευρώπη αυτή η δραστηριότητα δεν φτάνει ούτε καν το 8% του συνολικού όγκου συναλλαγών, σε άλλε περιοχές του κόσμου υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι αυτό το ποσοστό ξεπερνά 130% ήδη. Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μια σειρά κριτηρίων, προϋποθέσεων και ε, φραγμών που δεν επιτρέπουν μια ομοιογενή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ε, πούμε ότι έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες που δημιουργούν συνεχώς μια ανασφάλεια δικαίου και άρα έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Πρέπει λοιπόν να απλουστευτεί το νομικό πλαίσιο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και να υπάρξει ανάπτυξη και περισσότερη απασχολησιμότητα. Και οι καταναλωτές έχουν ενιαία νομοθεσία για τις ε, συναλλαγές που οδήγησε σε ανάπτυξη ε, του ψηφιακού εμπορίου και παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται του τομέα σε όλο τον κόσμο, οι ψηφιακές συναλλαγές την χάνουν κάποιες εχθρικής αντιμετώπισης. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, η δημιουργία θέσεων εργασίας ουσιαστικά εξαρτάται από τις μικρομισές επιχειρήσεις που στην Ευρώπη δημιουργούν 7 στις 10 θέσεις εργασίας. Μία μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να έχει την πολυτήλεια που μπορούν να έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές ε, να πολλά τα προϊόντα της ε, online, ε, μέσα στο διαδίκτυο και να πρέπει να προσαρμόζεται μέσω του διαδικτύου σε κάθε εθνική πραγματικότητα, εθνικό νομικό πλαίσιο, λογιστική πραγματικότητα ή ειδικέ διατάξει προ καταναλωτή. Συγκεκριμένο παράδειγμα, η ισπανική επιχείρηση Inditex, πολυεθνική εταιρεία, είναι, έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα πλέον, που ασχολείται με, τα, με την κλωστοφαντουργία. Και σύμφωνα με ισπανική εφημερίδα, αναγκάστηκε να επενδύσει 12 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυνατότητε που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία σε επιχειρήσεις μας είναι αναντήρητες. Τα τελευταία χρόνια για κάθε θέση εργασίας που χάθηκαν στην παραδοσιακή οικονομία, δημιουργήθηκαν 2,6 θέσει εργασία ε, στην ψηφιακή αγορά. Και αυτό είναι στοιχείο περίτρανο του, του πώ μπορεί η ψηφιακή αγορά να επηρεάσει θετικά για να μπορέσουμε να βγούμε την οικονομική κρίση. Και ιδίω αυτή την περίπτωση για να δημιουργήσει θέσει εργασία για του νέου, που είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο α, σταυροδρόμι. Θα μπορέσει να δημιουργήσει μια φιλική ή εχθρική τελικά αντιμετώπιση τη ψηφιακή οικονομία. Θα είμαστε στην προμετωπίδα ή θα είμαστε ο τελευταίο τροχός αμάξι σε αυτόν τον τομέα. Θέλουμε μια Ευρώπη χωρί φραγμούς ή θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε μια Ευρώπη που δεν θα δημιουργεί νέες θέσει εργασία. Αν οι επιχειρήσει μα δεν είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικέ σε άλλε. Ε, Τρίτε αγορέ, τότε η ιδέα της ενιαία αγοράς έναντι τη παραδοσιακή αγορά, δεν θα πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί πλήρως. Σήμερα έχουμε πια την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια ενιαία ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μάλλον επεξεργάστηκαν τελευταία διετία μια σειρά πρωτοβουλειών που θέτουν το πλαίσιο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος με τις διάφορες ανακοινώσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την, ε, το ψηφιακό θεματολόγιο, την πράξη για την ενιαία αγορά και τις διάφορες ομαδικές πράξεις που αφορούν ψηφιακή αγορά όπως ε, τα δικαιώματα του καταναλωτή κτλ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε διάφορες εκθέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και η ίδια η Επιτροπή μας εργάστηκε ε, εντατικά επί του θέματος και μάλιστα δημιουργήσαμε και μια ειδική της εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου εξετάζονται τα υφιστάμενα εμπόδια ε, και συγκεκριμένε καθαρές γραμμές που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση κατάστασης. Όμως, αναμφίβολα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, νομοθετικά μέτρα και θα πρέπει να αλλάξουμε άρδιν το παρόν σκηνικό. Συμφωνούμε όλοι ότι η καινοτομία είναι κλειδί στην όλη δυναμική ε, κατάσταση που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα. Και αυτή η καινοτομία είναι, ε, δεν είναι βιώσιμη αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και εμείς ιδίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν προκρίνουμε ένα ανοιχτό περιβάλλον που πραγματικά ευνοεί την ανταγωνιστικότητα. Τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα δεν επιτρέπουν στι επιχειρήσει μα να ανταγωνιστικούν επίση όρει όσου ε, ε, παρέχουν υπηρεσίε μέσω δικτύου. Αυτό αντίθετα ευνοεί αλλοδαπέ επιχειρήσει, κάτι που λειτουργεί βάρο των δικών μα επιχειρήσεων και ιδίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία σε όλο του το δυναμικό και όλο το δυναμικό που μπορεί να δώσει το ηλεκτρονικό εμπόριο για να μπορέσουν επίσης όρες να ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν εδρεωθεί ε, στο εμπόριο μέσω ίντερνετ. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να γίνει αυτό. Η ψηφιακή επανάσταση που έχει γίνει είναι η τάση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ιδάλλως θα μείνουμε πίσω και θα είμαστε πάλι ο τελευταίο τροχό στα Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν την επόμενη διετία θα κρίνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας μέσω μακροπρόθεσμα. Αν δεν γίνουν αυτές οι νομοθετικές αλλαγές, δεν θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα, πιστεύω, να υλοποιήσουμε με επιτυχία αυτές τις αλλαγές στο μέλλον. Αν δεν επιτύχουμε αυτό το στόχο κατά αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, φοβούμαι ότι θα έχουμε αποτύχει οι επιχειρήσεις που σήμερα είναι πρωτοπόροι στον κλάδο θα αποκτήσουν μια δεσπόζουσα θέση στο μέλλον. Και μέσα στην οικονομική κρίση δεν μπορεί η Ευρώπη να παραγνωρίσει αυτή την πρόκληση. Η έξοδος από την κρίση κατεμέ με, έχει ψηφιακή μορφή. Οι κατηρίε γραμμέ που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι πολλέ. Θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητε επιχειρήσει να χρησιμοποιούν το επιγραμμικό εμπόριο και ιδίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να άρουμε νομικά εμπόδια και ταυτόχρονα του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που να του επιτρέψουν να αναπτύξουν τι ε, συναλλαγέ του μέσω διαδικτύου όσο και πιο αποτελεσματικά. Π.χ. σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει νομιογενέ σύστημα ηλεκτρονική τιμολόγηση με ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική έγκριση να υπάρχει μεγαλύτερη διαθέσιμη πληροφόρηση για τις πωλήσει και τις δυνατότητες που παρέχει το μέσο, όπως και να υπάρχει μεγαλύτερη κατάρτιση μικρομεσαίε επιχειρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Να ενισχύσουμε πρωτοβουλίε προς το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο για την στήριξη του ηλεκτρονικού ε, εμπορίου ή ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τυποποίησης σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έπειτα, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα στη νέα ψηφιακή εποχή. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σίγουρα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά, επί της οποίας θα πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να πρικοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύστημα που να προστατεύει την ιδιωτική σφαίρα και να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, να αυξάνει την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ταυτόχρονα να δίνει επαρκή ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν την ηλεκτρονική τους δραστηριότητα χωρίς αυτό να σημαίνει ε, δυσβάσταχτο οικονομικό και διοικητικό άχθος. Η καλή ε, λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικές για τις εξαποστάσεως συναλλαγές. Η... Ένα από πραγματικό εμπόδιο το ε, διασυνοριακό εμπόριο είναι η αναγκαστική σωματική επαφή για την παράδοση προϊόντων. Παράγοντες που δεν επιτρέπουν μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να έχει διασυνοριακές συναλλαγές χωρίς δυσβάστακτο οικονομικό βάρος. Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των ήταν σίγουρα ένα άλμα προόδου ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη προστασία για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και θα πρέπει να ενσωματωθεί το των δυνατόν στις εθνικές νομοθεσίες. Παρά τα αυτά, υπάρχουν διάφορες πτυχές ε, του ζητήματος που θα πρέπει να εμβαθύνουμε για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή έναντι αυτού του μέσου. Οι πτυχές αυτές είναι, για παράδειγμα, η έγκριση ενός νέου κανονισμού για ε, τις εναλλακτικέ ε, μορφές επίλυσης ε, διαφορών online, ώστε να έχουμε ένα απλό αποτελεσματικό σύστημα για την επίλυση διαφορών μεταξύ αγοραστών και πολιτών. Επίσης χρειάζεται ένα κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει τις επιγραμμικές συναλλαγές. Επίσης να δοθούν πιο πολλοί πόροι στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προσοχής Καταναλωτή ώστε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ε, προστασίας καταναλωτή, κάτι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για προστασία καταναλωτή. Κατεμένει ένα μέτρο για την αύξηση της εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε εδώ να μιλήσουμε για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που πολλούνται μέσω διαδικτύου. Επίση, θα πρέπει να πλουστεύσουμε και να μηχανημίσουμε την νομοθεσία περί ΦΠΑ για τι επιγραμμικέ συναλλαγέ, ώστε να μειωθεί το διοικητικό άκθο, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να διακρίνουμε την επιβολή ε, ΦΠΑ για προϊόντα που ε, αγοράζονται ε, ηλεκτρονικά και να αναφέρομαι σε προϊόντα ε, με πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά Θα πρέπει να πλουστεύσουμε την κείμενη νομοθεσία, για παράδειγμα, σε θέματα διεθνής μεταχείρισης. Το άρθρο 25.2 της Οδηγίας Περιπηρεσιών είναι το περιβόητο άρθρο και έγινε πραγματικά περιβόητο λόγω της έλλειψης εφαρμογής του. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια για να το εφαρμόσουν. Τα πνευματικά δικαιώματα και η καταπολέμηση της πειρατείας είναι μεγάλες προκλήσεις. Σημαντικά ζητήματα με ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τη σχετική νομοθεσία περί υλοποίησης και διαχείρισης των δικαιωμάτων δημιουργού και να προσαρμοστούν στον 21ο αιώνα, να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ίντερνετ και να βελτιώσουμε τα συστήματα πληρωμών και να έχουμε πιο ασφαλείς πληρωμές μέσω του δικτύου, να έχουμε ένα νέο σύστημα λοιπόν, ε, που θα διέπει τις ευρωπαϊκές πληρωμές και περιμένουμε τη σχετική προσωπική επιτροπή ε, που θα ακολουθήσει τη στρατηγική η οποία ήδη ανακοινώθηκε. Σε γενικές γραμμές, Αυτές είναι οι γενικές γραμμές δράσης που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υλοποιηθούν. υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που δεν έχω το χρόνο να αναφέρω. Αλλά αναμφίβολα θα ήθελα να συμπεριληφθούν. θα ήθελα να ακούσω βεβαίω πρώτα απ' όλα τι γνώμε των συναδέλφων εδώ στην Επιτροπή μα για να καταλάβω ποιε είναι οι προτάσει του. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω επί του θέματος. Δεν αναφέρθηκα στο e-commerce, το οποίο είναι ζωτική σημασίας και θα αναφέρεται στην έκθεση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω. Θέλω να ακούσω τις γνώμες των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Good. Uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεξοδικότατη παρουσίαση. Ας ακούσουμε τώρα τους Κιώδης και όποιον άλλον θα ήθελε το λόγο. Ε, ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος, ο κύριος Λούχε Γκάρντεν, ο κύριος Μάντες, ο κύριος Έγκστρομ είναι εδώ, κύριε Μακλάρκιν, Γκούσταυσον από την ΚΟΕ δεν είναι εδώ η κυρία Λαμάτης από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΚΤ. Θα σας ακούσουμε στη συνέχεια. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτε έχει ήδη πει ότι θέλει να μιλήσει. Ε, δίποτε άλλος θα μου κάνει ένα σήμα. Ας αρχίσουμε με τον καθηγητή Κορέιντε Κάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα για λίγα δευτερόλεπτα να ποτίσω φόρο τιμή σε έναν βουλευτή, τον Μίγκελ Πόρτας, που απεβίωσε στα 53 έτη του εχθές. Είναι θλιβερό για τον συμπατριώτη, φίλο, βουλευτή, πεπισμένο ευρωπαϊστή και παρόλες τις ιδεολογικές ε, διαφορές πραγματικά ε, ήταν κάποιος που χαρακτηριζόταν από μεγάλη αφοσίωση. Αυτά. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρία Σεσεβάρια Εσεβερία, συγγνώμη, για τα όσα έκανε στην Επιτροπή μας, για αυτή την έκθεση. Ανέκαθεν ήταν η ψυχή της εργασίας για αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι σήμερα έχουν ε, ε, τα πράγματα δυσκολέψει και είναι πολύ πιο δύσκολα ε, από ό,τι περιμέναμε στην αρχή. Πριν από ένα χρόνο νομίζαμε ότι είναι εύκολοι οι υπολογισμοί και ότι είναι ένα μαθηματικό ζήτημα. Μιλούσαμε για τα ποσοστά και θεωρούσαμε ότι είναι με μηχανικό τρόπο εύκολο να αυξήσουμε τον αριθμό των συναλλαγών Βλέπουμε όμως ε, πόσο δύσκολη αποδεικνύεται ε, αυτή η κατάσταση και πόσο δύσκολο είναι να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό, τους φραγμούς, ε, ε, την ε, δυσαρέσκεια των καταναλωτών, την έλλειψη κατανόηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον κατακαιρματισμό που ισχύει στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργού. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, τους διαφορετικούς φόρους προστιθέμενη αξία, τα διαφορετικά συστήματα επιγραμμικής πληρωμή. Ε, το θέμα διανομής, ε, ε, το θέμα διευθέτησης των διαφορών, προστασίας των δεδομένων, όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται και προκύπτουν, θα έλεγα, αντιευρωπαϊκές καταστάσεις, δηλαδή διακριτική μεταχείριση λόγω εθνικότητα, όταν κάποιο αγοράζει διαδικτυακά στη συνέχεια ή στο σελίδες ε, όπου δεν υπάρχουν ε, επαρκή δεδομένα για τις διασυνοριακές ε, συναλλαγές ούτω ώστε ο καταναλωτής να έχει πλήρη ενημέρωση και να έχει το δικαίωμα επιλογής. Επίσης δεν ξέρουμε πάντοτε ποιο είναι ο συνομιλητής μας, το άλλο συμβαλόμενο Στι μέρος ε, στις επιγραμμικές ε, πωλήσει. Πολλά προβλήματα βλέπουμε, όλα τα εμπόδια, όλους τους φραγμούς ε, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιστορική αγορά και καταλαβαίνετε ότι αυτό πλήττει την οικονομία, την καινοτομία, την απασχόληση κυρίως των νέων, όπως τόνισε ο κύριος Δεσεβάρια και άρα ε, δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας προσφέρεται τώρα. Μας παρουσιάζει μια πολύ λογική ανακοίνωση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εύστοχες, ε, πρόσφορες προτάσεις, με, με μερικές συμφωνούμε. Η ομάδα εργασίας μας ήταν ήταν εξαιρετικά χρήσιμη στο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς. Η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, κυρίως όταν μιλάμε για τις αγορές, είναι μια συνενετική διαδικασία. Ε, στην ομάδα εργασίας ε, τι κάναμε σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάντοτε υπεραμηθήκαμε τις θέσεις μας και θέλαμε να προχωρούμε με σταθερό τρόπο Βρισκόμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με όλες αυτές τις δυσκολίες ε, παρόλα αυτά που φανταζόμασταν στην αρχή και ε, θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο του Πάμπλο Άριας ε, Εσεβάρια θα συμβάλλει τα μάλλα στην μεταξέλιξη, την περαιτέρω ανάπτυξη αν θέλει, της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστούμε κύριε Κορέα. Ο κύριος Έγκστρομ τώρα. Thank you. Um, Συμφωνώ με αυτά που είπαν ε, πολλοί προλαλήσαντες και με αυτά τα οποία λέει στην ανακοίνωσή της η συγκήτρια ε, αλλά πρέπει να πούμε ότι η, ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι αυτό που μας απασχολεί και θέλουμε να προωθήσουμε και η ψηφιακή αγορά θα είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτή την ε, ε, κατά πρωτοβουλία έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, αν κοιτάξουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, όλοι συμφωνούμε ότι ε, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο σαν πολιτική μπορούμε να υπαγορεύσουμε εκ των άνω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε, αλλά πρέπει να αυξήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και αν έχουμε την ε, ίδια ε, νομοθεσία για τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη θα ε, αρχίσουν ε, οι καταναλωτές ε, να αγοράζουν από τη χώρα τους αντί από ξένες χώρες. Αλλά πρέπει να δούμε γιατί ήδη έχουμε αποφασίσει κατά της εναρμονήσεως. Υπάρχει λοιπόν μία συνέπεια εκεί και όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφερόμαστε σε παρτίδες και πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, διότι πέραν της ανησυχίας ότι δεν θα παραδοθεί το υλικό και ούτω καθεξής υπάρχει ο κίνδυνος τώρα ε, για τα τελωνία να κατάσχουν ε, τα προϊόντα που αγόρασαν για λόγους τελείως ακατανόητες για τους καταναλωτές. Άπαξ και ε, η νομοθεσία δίνει αυτό το δικαίωμα στα τελωνία. Ε, αγοράζω κάτι από το εξωτερικό, είτε από την Αμερική από ένα άλλο κράτος μέρος. Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβαιναν ποια είναι η διαφορά. Ε, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την οδηγία που εφαρμόζεται στα τελωνία, ε, εάν υπάρχει ταινία ε, μπορεί η ταινία αυτή να κατασχεθεί διότι υπάρχει μία διαμάχη πνευματικών δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο αντικείμενο και αυτό που θα γίνει είναι ότι το άτομο που εμπλέκεται θα νευριάσει, θα το πει σε όλους τους φίλους του και θα πει ότι ουσιαστικά δεν, δεν πρέπει κανείς να εμπιστεύεται και να αγοράζει κάτι στο εξωτερικό. Υπάρχει λοιπόν εκεί μια συνέπεια μεταξύ των καλών επιχειρημάτων που έχουμε στην αρχή και κάτι άλλο που κάνουμε σε πολλά νομοθετικά θέματα. Επίσης όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές στο διαδίκτυο πιστεύω ότι όλοι θα θέλαμε να υπάρχουν περισσότερες ένομες εμπορικές προσφορές για αυτούς που θέλουν να πληρώσουν για τα πολιτιστικά αγαθά και να αγοράσουν οτιδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν χώρες οι οποίες προσπαθούν να σας προσφέρουν υπηρεσίες και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πρόθυμος να αγοράσει μουσική παραδείγματος χάρη αλλά ε, ε, υπήρχε η δυνατότητα αυτή σε 7 από τις 27 χώρες. Όχι γιατί οι άλλες χώρες δεν θέλουν, αλλά πρέπει να ε, διαπραγματευτούν με την οργάνωση που διαπραγματεύεται τα πνευματικά δικαιώματα σε κάθε χώρα η οποία ε, διαπραγματεύεται τα πνευματικά δικαιώματα και με τις, ε, τους πολλαπλασιασμούς πρόκειται για 157 διαπραγματεύσεις που είναι κάτι που δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε κάποιος ε, τρόπος θα πρέπει να υπάρχει για ένα ευρωπαϊκό για μια ευρωπαϊκή κατοχήρωση των πνευματικών δικαιωμάτων ε, και κάτι θα πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ορισμένα κατοχυρωμένα συμφέροντα θα ζημιωθούν. Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε το θέμα αυτό, πολύ φοβάμαι ότι εγώ δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξο, διότι βλέπουμε τι γίνεται και ίσως υπάρχει κάποιος τρόπος να λύσουμε τα θέματα αυτά μέσω της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα μας στείλει μία πρόταση σύντομα. Δεν θα έρθει άμεσα και κατευθείαν στην Επιτροπή μας, αλλά κάποια ώρα θα φτάσει. Κυρία Μακλάκη. Ευχαριστώ και καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση του επί του θέματος και θα έλεγα την εντυπωσιακή ομάδα θεμάτων που έθεσε στην ομάδα εργασίας. Να πούμε ότι 2,63 ευρώ είναι γενικότερη γενικότερη εργασιών στον τομέα και σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό επί κατά 100 αν θέσουμε το κατάλληλο πλαίσιο. μελέτες λένε ότι σύντομα θα έχουμε 3 δισεκατομμύρια ε, πολίτες ε, online και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε. Λοιπόν, αν μπορέσουμε να δράξουμε πλήρω τα ωφέλη από την ψηφιακή αγορά, πραγματικά θα ήταν κάτι εξαιρετικό. Γιατί υπάρχει τεράστιο δυναμικό και πρέπει να το καταλαβαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε λοιπόν ε, σύντομα να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλε τι προτάσει που μα έχει υποσχεθεί. Πρόταση κλειδί ειδικά για το πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείριση αυτών, για το copyright. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευέλικτο σύστημα διοδότησης, προστατεύοντα ταυτόχρονα τα δικαιώματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών για να υπάρχει πραγματικό όφελος για του καταναλωτέ. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο αν απλουστεύσουμε τι διαδικασίε ε, εδαφικού συστήματο αδειοδότηση και αν εσυγχρονιστούν τα σχετικά εθνικά συστήματα. Και, γιατί αυτή τη στιγμή η νομοθεσία πνευματική ιδιοκτησία είναι πάρα πολύ περιπλοκή και δεν δίνει όλα τα ωφέλη στου καταναλωτέ. Τώρα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε αντιμετωπίζουν του περισσότερου φραγμού ε, και εμποδίζει αυτό την ανάπτυξή του σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η κείμενη νομοθεσία. Είναι γι' αυτό κομμάτι της ολοκλήρωσης της ενίας ψυχικής ώρας. Και θα πρέπει να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε τη διασυνοριακή και επιγραμμική δραστηριότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Και να αναφέρω ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση, διασύνδεση των πολιτών με τι προμεσαίε επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα απ' όλα να απτύξουμε τις ευρυζωνικέ υπηρεσίε πριν ανοίξουμε την και αγορά στου πολίτε. Θα πρέπει επίση να δούμε πώ ε, θα ε, επιλύσουμε το θέμα τη επίλυση διαφορών των καταγγελιών διασυνοριακό και και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση για το μηχανισμό επιγραμμικής επίλυσης διαφορών που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ε, που θα διέπει τις ε, διασυνοριακές πληρωμές. Από εκεί και πέρα συμφωνώ με την πρόταση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για την ε, υλοποίηση του συνεργασία μαζί με τα κράτη-μέλη, μέσω και του IMI. Τώρα, για τις προτάσεις που ζήτησε ο εισηγητής, θεωρώ και εγώ προτάσεις με σαφή ευρωπαϊκή προσεθέμενη αξία. Συμφωνώ και εγώ. Όμως, ε, διαφωνώ με μία πρόταση, με ένα sales board που εμπεριέχει πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας πείσετε εμάς εδώ θέτοντας το επιχείρημα ότι 27 διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες δημιουργούν πρόβλημα. Αυτό είναι σίγουρα το θέμα. Είναι να εστιάσουμε περισσότερο σε πρακτικές λύσεις. Ίσως χρειάζεται κωδικοποίηση πολύ απλά όσων ήδη έχουμε θετήσει με τα δικαιώματα του καταναλωτή και στην οδηγία, αντί να δημιουργήσουμε ένα εντελώς καινούριο και πολύ δαπανηρό σύστημα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Παρακαλώ τον εισηγητή και του συναδέλφου, να είμαστε πολύ λογικοί στον τρόπο που προτείνουμε να δαπανίσουμε το χρήμα των Ευρωπαίων ε, φορολογουμένων. Πρέπει λοιπόν πέρα από τα λόγια να μπούμε σε πράξεις για να έχουμε πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Uh, thank you very much, Mr. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω θα περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Ε, να σας πω ποιοι είναι εδώ. Mrs. Mrs. Gallo Υπάρχει κάποιος άλλος θέλει να εγγραφεί στον κατάλογο ομιλητών. Όχι, η κυρία Κορατσαμπίλτ. Ευχαριστώ, Μάλκον. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτέλους είναι πολιτική προτεραιότητα το να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Είναι η ώρα των σοσιαλιστών και μας λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν χρήματα που δεν υπάρχουν. Εξαπατούν τους καταναλωτές, υπόσχονται ανάπτυξη με χρήματα όμως που δεν υπάρχουν για να δαπανηθούν. Και εμείς ε, αντιπροτείνουμε να απελευθερώσουμε τον εκμετάλλευτο δυναμικό της αγοράς. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέθεσε πρόταση με 16 συγκεκριμένες δράσεις για το οδικό χαρτί. Αναφέρομαι στο φίλο από το ΕΛΚΑ. Ε, ε, πρόκειται για την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη δεν μπορεί κανείς να τη δημιουργήσει του μειόντος. Θα πρέπει να άρουμε τα προσκόμματα, τους φραγμούς που υπάρχουν, να, να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της κίνησης στο διαδίκτυο, όπως έχουμε ήδη καταφέρει στην εσωτερική αγορά. Δεν μπορεί αυτά να ξεκινήσουν από την κορυφή προς τα κάτω. Εδώ και δύο χρόνια εργαζόμαστε εντατικά ούτως ώστε να επιτύχουμε εναρμόνιση των κανόνων της προστασίας του καταναλωτή. Εσείς που ήσασταν όλο αυτό τον καιρό όταν εμείς αγωνιζόμασταν, γιατί παραπονιέστε τώρα, μα που ήσασταν, τι κάνατε, αγωνιστήκατε εσείς για την εναρμόνιση. Όχι, λέτε ότι προτού καν λάβετε την πρόταση δεν, θα δεν την εμπιστεύεστε. Για πρώτη φορά συζητάμε την έκθεση και λέτε σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Τι στο διάβολο θέλετε επιτέλους, δώστε μας και κάποιες εναλλακτικέ ε, λύσεις. Ε, ε, πώς θα επιτύχουμε την ψηφιακή εσωτερική αγορά και για τη Σουηδία και για την Ευρώπη. Αντί να παραπονιέστε και να αντιλέγετε σε όλα και να τους κατακρίνετε όλους, κάντε κάτι. Ε, θα ήθελα τώρα να σχολιάσω δύο σημεία σε αυτή την εξαιρετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δράση υπαριθμών 3. Ε, χαίρομαι που ε, θίγει το ζήτημα των θεμητών όρων ανταγωνισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το B2B από την επιχείρηση σε επιχείρηση, τις συναλλαγές από επιχείρηση προς ιδιώτες, πολύ θετικά όλα αυτά. Μιλάμε για κώδικα διοντολογίας, μιλάμε για τα εφαρμοστικά μέτρα, ε, μετά από αυτήν την έκθεση που αναφέρατε για την δικαιότερη εσωτερική αγορά στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θέλει να κρατήσει συνοχή σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Για τη δράση παριθμών 5 χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για σύγκριση ε, όχι μόνο των τιμών αλλά και της ποιότητας ε, των προϊόντων. Αυτό το επιδιώκουμε εδώ και καιρό, κυρίως τη Λιανική για τα τρόφιμα ούτω ώστε να καταβάλουμε το τίμημα, αλλά να έχουμε και την αντίστοιχη ποιότητα. Τι εννοεί ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να επεκταθεί λίγο. Είναι εξαιρετικά περίεκτική αυτή η πρόταση, γιατί καλείται να ευρύτατο φάσμα ενίσχυση υποδομή μέχρι και το ε, να αποκτήσει ο καταναλωτή ε, περισσότερε εξουσίε σε σχέση με το ραδιοφάσμα, την κατανομή του ραδιοφάσματο, οι καταναλωτέ να βρίσκονται σε μια καλύτερη θέση. Ωραία, συνεκτικό είναι το πλαίσιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώ ακριβώ ε, θα έχει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση για να καταργήσει όλους τους περιορισμούς ε, και να ε, παλέψει με τα κράτη-μέλη που ακόμη αντιστέκονται για την καθίδρυση μια ψηφιακή εσωτερική αγορά. Ευχαριστούμε κυρία Κορατσαμπίλτ. Η κυρία Μπαχαέρ. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο ήδη έχει θυγεί και αυτό είναι το σημείο τομής μεταξύ της ε, ψηφιακής αγοράς, της ουσιαστικής αγοράς, ε, της παραδόσεως, ε, της επιστροφής. Έχουμε διάφορες πτυχές της ενιαίας αγοράς, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο, στην παράδοση, στον έλεγχο ή στην εφαρμογή οι μεταφορικές εταιρείες είναι ένα αδύνατος κρίκος, το κόστος της μεταφοράς είναι ένα δύνατο σημείο, πρέπει να υπάρξουν διακινήσεις μεταξύ λογαριασμών και αυτό είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι προσπαθούν να εισέλθουν στο χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν δυνατότητες να εκπαιρεωθεί μία πληρωμή αλλά υπάρχουν και ιδιομορφίες και ιδίως όσον αφορά του όρου πληρωμής, το δικαίωμα επιστροφής, ε, τα δικαιώματα του καταναλωτή ε, και άλλα παρεμφερή χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσπάθεια για ενίσχυση των θεμάτων διότι έχουμε δυνατότητες αναπτύξεως πέραν του 80% ε, και δεν τα έχουμε ε, υλοποιήσει στην πραγματική πώληση αλλά βάσει μιας μελέτης την οποία είδα μπορεί να δημιουργηθούν 35.000 νέες θέσεις εργασίας στα πλαίσια της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Είναι πάρα πολλά άτομα που μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και μπορούν να προκαλέσουν ποσοστά αυξήσεως αλλά δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Ε, μια Ευρώπη που δεν έχει λεφτά στην τσέπη της δεν θα ξοδέψει. Οπότε με την ενίσχυση της ψηφιακής αγοράς και του ψηφιακού εμπορίου μπορούμε να μειώσουμε ε, το πραγματικό εμπόριο, ιδίως στην Ήπεθρο όπου η ε, υποδομή ε, των δικτύων ε, είναι ανεπαρκής. Ξέρουμε ότι υπάρχει μία συγκέντρωση σε εμπορικά κέντρα όπου είναι δύσκολο να υπάρξει παρακολούθηση και ο χώρος αυτός αντικαθίσταται από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι με την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου αυτές οι επιπτώσεις θα ενισχυθούν Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την ύπεθρο αλλά για να μην την αποκόψουμε από το ηλεκτρονικό εμπόριο επανερχόμαστε εις την ανάπτυξη των δεικνύων στις ευρυζωνικές συνδέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί αν θέλουμε να υπάρχει μία μετατόπιση προς την ψηφιακή ψηφιακή αγορά προς το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. κυρία Καλάορο, ο κύριος Σβάμπ και μετά ο κύριος Έγκστρομ στο τέλος και η κυρία Κοράτσα Μπίλ θα ήθελα να ακούσει τα σχόλιά σας. Η κυρία Κάλλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τον υποστηρίζω πλήρως και θα συνεργαστώ μαζί του όταν ε, και όσο χρειαστεί. Σε αυτή τη συζήτηση ασχοληθήκαμε με τα δικαιώματα δημιουργού ακούσαμε και την παρουσίαση του συναδέλφου Έγκστρομ, προσπαθεί να μας πείσει, παραδείγματο χάρη, ότι θα πάρουμε ένα τηλέφωνο εκεί στα σύνορα, ενώ ξέρουμε ότι αποκλείονται οι προσωπικές ε, χειραποσκευές. Ε, ήθελα μόνο να σας πω ότι για τα ψηφιακά προϊόντα και το ΦΠΑ, εφόσον θέλει να είναι νόμιμη, προσβάσιμη και φτηνή θα έλεγα η προσφορά, ε, θα ήθελα να υποστηρίξει την πρότασή μου τότε, αυτό που δεν έγινε από πλευρά των Πρασίνων. Χαίρομαι λοιπόν ε, και τα λέω αυτά πρωτού ξαναπάρει το λόγο γιατί θέλω να ακούσω τι πιστεύει για την έκθεσή μου. Θα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση σχετικά με το ότι για το 2012 μας έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος, το cloud computing. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και συσχετίζεται με αυτό που συζητούμε, διότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό για την αύξηση του αριθμού θέσεων απασχόλησης και ένα πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ακριβώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί εκείνες είναι που δεν έχουν συνήθως τους πόρους για να επενδύσουν στις τεχνολογίες εχμής έξω και η παρατήρησή μου, γι' αυτό εφιστώ την προσοχή σας αυτό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Well, thank you, Mrs. I... Σας ευχαριστούμε. Καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι τη γνωμοδότησή σας για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών θα, τη συζητήσουμε αργότερα γιατί όντως χρειαζόμαστε υψηλότερη ποιότητα για να κινητοποιηθούμε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μέσα στην εσωτερική αγορά. Κύριο Σφάπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ελέγχθησαν οπότε εγώ θα περιοριστώ σε παρατηρήσεις που μου φαίνεται ότι είναι βασικό να τονίσω. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ με την οριζόντιο στρατηγική του προσπαθεί ε, ε, ε, προωθήσει την εσωτερική αγορά και να τη διαμορφώσει όπως άλλωστε και την ηλεκτρονική αγορά με διάφορους τρόπους όπως η σημερινή ε, νομοθεσία ε, που ακόμη ε, δεν προσδίδουν στην Ευρώπη και στον καταναλωτή την ποιότητα την οποία επιθυμούμε για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε. Οπότε αυτό ανησυχεί τους ε, καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν διασυνοριακά. Ευχαριστώ τον κύριο Αρίας που εξέταξε το Ευρωβαρόμετρο όπου λέγεται ότι πολλοί ξεκινούν να κάνουν ε, ε, αγορές διασυνοριακές αλλά στο τέλος δεν τους παραδίδουν είτε διότι δεν μπορούν μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία της της ε, πιστοτική τους κάρτας διότι τα συστήματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι εντός της χώρας και για ένα σωρό άλλες παραμέτρους που και πολύ σωστά το είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλντ ε, δεν καλύπτονται από το γεγονός απλώς ότι υπάρχει έλλειψη, ε, έλλειψη αξιοπιστίας αλλά πρέπει να υπάρχει μία εξέλιξη στην οποία η Κομισιόν θα εμπλακεί θετικά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να επανέλθω εις ε, την στολή που έγραψε ο πρόεδρος της Επιτροπής ής ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά για να επηρεαστεί θετικά και η ε, ψηφιακή οικονομία αλλά υπάρχουν κανόνες οποίους γενικότερα έχουμε χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη. Ο κύριος Έγκστρομ, νομίζω ότι και εσείς έχετε λόγο να απαντήσετε. Κύριε Κορατσαπίλ, και και κύριε Καλαρ, παρότι που έφυγε, θέλω να απαντήσω και στις δύο συναδέλφους. Είμαι πολιτικός, αλλά δεν ισχυρίζομαι ότι μπορώ να προσφέρω απτές λύσεις για κάθε πρόβλημα. Ίσως να μην είμαι πολιτικός 100% ακόμη. Όταν μιλούμε για το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, θα έλεγα να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, μήπως κάνουμε και λάθος. Ας δούμε και πάλι το ίδιο θέμα. Πάντοτε υπό το φως και αυτής της έκθεσης και όλων των λοιπόν πρωτοβουλειών για την πρόθεση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και έχει δίκιο ότι λείπουν κάποια πράγματα από, αυτό το κανονισμό, από τον κανονισμό, αλλά δεν ε, σημαίνει ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή και ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται κανείς να μεταβεί πρακτικά. Οπότε δεν τίθεται αυτό το θέμα των χειραποσκευών, όπως ακριβώς το θέσατε. Σε ό,τι αφορά τώρα το copyright και την ε, ψηφιακή αγορά, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Να σας πω ότι χθες ε, και εγώ παρουσίασα, δημοσίευσα ένα βιβλίο ακριβώς για το θέμα του copyright, το οποίο διανύμα σήμερα σε όλους τους συναδέλφους, θα το βρείτε ε, αν θέλετε ε, εκεί που παίρνετε τη σας. Και θα δείτε ποια είναι η άποψή μου για το ζήτημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες κοινωνίες που πραγματικά επηρεάζουν ε, τα πράγματα μέσω των δικαιωμάτων νομικής ιδιοκτησίας και μας κρατούν, θα έλεγα, πίσω από την πλήρη ολοκλήρωση ψηφιακή αγοράς. Σε κάθε περίπτωση προσβλέπω συνεργασία με όλους σας για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, λοιπόν Εγώ θα σας δώσω μια πλατφόρμα για να λανσάρετε το βιβλίο σας και με χαρά να το διαβάσουμε όλοι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, αλλά αν κάνουμε μια γνωμοδότηση ε, για αυτό το ζήτημα, έτσι θα μπορούσαμε να το δούμε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αν μπορούσα να κάνω κι εγώ κάποια λίγα σχόλια επί του θέματος. Συμφωνώ με τους συναδέλφους πρώτα απ' όλα ότι το έγγραφο της ΓΔΜ είναι ένα πολύ καλό κείμενο, ένα εμπεριστατωμένο κείμενο και ήδη στην Επιτροπή μας και σε άλλες επιτροπές τρέχουν παράλληλα διάφορα σχετικά ζητήματα. Ο κύριος Αρίας τα ανέφερε. Οπότε πρέπει να εστιάσουμε πιο πολύ στα κενά που πρέπει να καλύψουμε. Υπ' αυτή την έννοια, να επαναλάβω αυτό που είπε και η κυρία Κορέτσα Πίλτ. Πρέπει να δούμε το θέμα τον, ε, που προβλέπει ο ανταγωνισμός και το δίκαιο περί ανταγωνισμού και ε, ίσως να μην είσαστε απόλυτα σαφείς και μεριτές πρωτοβουλίες εν προκειμένου. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι το διαδίκτυο μπορεί να προωθήσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα. Και δίκιο έχει και η Επιτροπή όταν επισημαίνει κάποια δυνητικά προβλήματα που μπορούν να ανακύπτουν όταν υπάρχει τεράστια γκάμα επιλογών. Και το θέμα πολύ συχνά είναι πώς μπορεί κανείς να βρει γνήσια ανεξάρτητες πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι όλων. Οπότε το θέμα της διαφάνειας. Πραγματικά κρίσιμο ζήτημα αυτό. Κάτι άλλο τώρα που ήθελα ιδιαίτερα να θέσω αφορά κάτι που έθεσε η κυρία Μακλάρκεν για τα δικαιώματα του καταναλωτή, γενικότερα τα θέματα του καταναλωτή. Με ενδιαφέρον παρατήρησα ότι στο εγγραφό της η Κομισιόν, και θα αναφέρω εδώ, λέει ότι για το 2012, αν, ουσιαστικά 22 Μαΐου συγκεκριμένα, αυτή την πληροφορία που λάβαμε από το γραφείο του κ. Ντάλι ότι θα μας προσθέσει η Κομισιόν την ε, Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καταναλωτή. Και σίγουρα αυτό που θα επηρεάσει τα μάλα της συμπεριφορά του καταναλωτή είναι η ψηφιακή αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε αυτές τις προτάσεις. Υπ' αυτή την έννοια να αναφέρω στην μια συνάντηση με τον κύριο Αρά στην ομάδα εργασία είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από, την, από το Ευρωπαϊκό και το καθηγητή. και ότι είναι καλό να υπάρχει μια σύμβαση πλαίσιο που θα χρησιμοποιείται στις επιγραμμικές συναλλαγές ένα πολύ απλό έντυπο. Αυτό ουσιαστικά που είπε η κυρία Κλάρκν. Δηλαδή, πολύ απλό έντυπο που θα λαμβάνει υπόψη τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή σε κάποια στοιχεία. Κατά με αυτή η λύση Μα δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες να προχωρήσουμε μπροστά παρά ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πολίσεων. Γιατί βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη είναι απρόθυμα να κινηθούν προς αυτήν την κατάσταση. Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε γρήγορα σε πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων καταναλωτή στο διαδίκτυο, αυτή η πρόταση καλό είναι να αναφερθεί. Και νομίζω ότι και η πρόταση του κυρίου Αρίας είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για να κινηθούμε ε, κατά, ε, παράλληλα. Παράλληλα με ό,τι προβλέπει η πρόταση νομοθεσίας ε, για τις πωλήσει. Τώρα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή στην κυρία Λαμότα, αν θέλει να απαντήσει εντάχει στη συζήτηση και μετά θα κλείσει η συζήτηση ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Αρχίζοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία την συνεργασία με τον κύριο Αρία Σεβάρια και την πολιτική του ομάδα που εδώ και 1,5 χρόνο θέτει το ζήτημα επιτάπητος και μας επιτρέπει έτσι να συζητήσουμε τα επιμέρους ζητήματα. Ε, στα πλαίσια λοιπόν των εργασιών της ομάδας εργασίας και μετά την δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη σήμερα διαπιστώνουμε μια μεγάλη σύγκληση απόψεων για την ανάγκη να δράσουμε ταχύτατα, ώστε να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά, ε, δοθήσεις και της επίπτωσης της, επί της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πράγμα που χρειαζόμαστε διακάως. Ε, ως προς την διαπίστωση και ως προς το σχέδιο δράσης ε, βλέπω ότι υπάρχει σύγκληση απόψε ακόμη και με το Συμβούλιο. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ε, έκανα, παρευρέθη σε μια πρώτη συζήτηση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου σε σχέση με την ανακοίνωσή μας. Η δεύτερη συνεδρίαση εκτελήσεται τώρα παράλληλα σήμερα το πρωί. Ε, πάντως ε, από την πρώτη συνεδρία ήταν θετικά ε, τα αποτελέσματα. Βεβαίω ο διάβολο στη λεπτομέρεια κρύβεται, οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώς τι διάφορε προτάσει για να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενίας αγοράς, ούτε καν μια συλλογική ενία δράση που θα μπορούσαμε να προαγάγουμε και να διαπραγματευτούμε. Πρόκειται μάλλον για μια δέσμη δράσεων που σχολιάστηκε εκτενώς στη σημερινή συζήτηση και εκτιμούμε τη σημασία που αποδίδεται στις υποδομές, κυρίως στην Ήπεθρο, ε, τα θέματα ανταγωνισμού που επίσης δονήσαμε στην ανακοίνωσή μας, ε, παραδείγματος χάρη αυστηρή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με τους τους περιορισμούς. Όταν μιλάμε για αυστηρότητα σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση γιατί ενδέχεται να σημειωθούν και καταχρήσεις. Εν παρόδο να πω στην κυρία Κορέτσα Μπίλτ ότι ναι, ε, έχουμε κατά νου και συνυπολογίζουμε και την έκθεση για, την για το λιανικό εμπόριο το 2010, αν θυμάμαι καλά, και η δράση 3 συγκεκριμένα σχετίζεται με τις συναλλαγές B2B από επιχείρηση σε επιχείρηση και με την κυρία Λαζάροβα, ούτω ή άλλω και του συναδέλφου τη. Είχατε στο παρελθόν την ευκαιρία να συζητήσετε αυτό το θέμα. Ε, κατόπιν ενημέρωση και δικαιώματα δημιουργού. Ε, όταν λάβουμε το σύνολο των προτάσεων θα τοποθετηθούμε, αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια συμφωνία για να σημειωθεί πρόοδο στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο που αναφέρεται στην ανακοίνωσή μα και καλό είναι να το ε, έχουμε διαρκώ κατά νου. Όταν λοιπόν διαπραγματευόμαστε νέες προτάσεις, πάντοτε πρέπει να ε, έχουμε κατά νου την ψηφιακή επίπτωση των ε, νέων δράσεων. Αυτό ε, αναφέρεται και στην αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί περιγράφονται κατευθυντήριες γραμμές. Όλες οι νέες νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ε, Συν το χρόνο θα επανέλθουμε σε όλες αυτές τις επιμέρους προτάσεις ε, και είμαστε στη διάθεση του κυρίου Σεβαρή αν χρειάζεται βοήθεια για τη συνέχιση των εργασιών του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι και το Συμβούλιο σταδιακά σημειώνει κάποια πρόοδο, διότι είναι ε, ε, σημαντική προτεραιότητα για μας αυτό το θέμα. Η κυρία Γκέπχαρτ απουσίαζε αλλά θέλω να την ακούσουμε γιατί ήταν και εκείνη στην ε, συνεδρίαση της ΚΟΖΑ και εφόσον πραγματευτήκαμε θέματα ενίας αγοράς, ε, ακούσατε και την κυρία Κρούς που παρουσίασε την, το σχέδιο για την ενιαία αγορά. Είναι πολύ καλό που συνιστά το θέμα προτεραιότητα για όλους. Ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι σχέση με αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ήταν όντω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση εχθές το πρωί στην Κοπενχάγη για την ψηφιακή αγορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς επιθυμεί να προβεί σε πολύ προοδευτικέ εργασίες τι οποίες χαιρετίζουμε. Ήταν καλό να δούμε ότι μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων υπήρχε μεγάλη συνένεση και ε, καλύψαμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή όντως ήταν ε, μια εξαιρετική εργασία σχεδόν τριών ωρών και πιστεύω ότι θα υπάρξει και μία γραπτή ενημέρωση για τα πορίσματα που θα καταρτιστεί από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε στη σωστή οδό και γενικώ χαιρετίστηκε πάρα πολύ ό,τι έχει επιτευχθεί σε αυτό το τομέα. Κύριε Αρία, θα θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση και δίνοντας ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω κάτι στον κύριο Πόρτας. Εγώ δεν γνώριζα ότι αποβίωσε χθε ο Μίγκελ Πόρτας. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη για αυτή την επενθύμηση. Να απευθύνω το θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Τους άκουσα με μεγάλη προσοχή. Θεωρώ ότι κινούμεθα στην ίδια κατεύθυνση όλοι. Και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης. Υπάρχουν και πράγματα που δεν αναφέραμε πριν, όπως είναι η πρόσβαση της υπαίθρου στο ηλεκτρονικό επόριο, η χρήση του φάσματος και η πρόσβαση ε, των αγροτικών περιοχών στο φάσμα είναι ζητήματα που θα λάβω υπόψη και θα είναι πραγματικά παρόντα στο κείμενό μου. Τώρα, κάτι που ήλθε και επανήλθε στη συζήτηση και συμφωνούμε όλοι επ' αυτού είναι η απλούστευση της κειμένης νομοθεσίας. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί για την ανάπτυξη όχι μόνο του ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι αυτή τη στιγμή προς ζήτηση, αλλά γενικότερα. Έτσι πιστεύω ότι απαντώ σε διάφορα από τα ερωτήματα που ακούστηκαν στη συζήτηση. Για πρώτη φορά ε, πνέει ούριος άνεμος, θα έλεγα, στα θεσμικά όργανα. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να συμφωνήσουμε τώρα σχετικά με το πώς θα το κάνουμε. Αλλά θέλουμε πιο πολύ Ευρώπη σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, για το χρονοδιάγραμμα να πω λίγα λόγια. εξέταση του σχεδίου έκθεσης στις 20 Ιουνίου. Καταλεκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών η 10η Ιουλίου, εξέταση τροπολογιών στις 18 Σεπτεμβρίου, διαπραγμάτευση για το συμβασμό επιτροπολογιών στις 10 Οκτωβρίου, τελική προθεσμία, και στις 11 Οκτωβρίου συνάντηση με την Επιτροπή και αν όλα πάνε καλά να περάσει η έκθεση από την Ολομέλεια το Νοέμβριο. Ελπίζω να μην έκανα κάποιο λάθος, αλλά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Αυτές είναι οι ημερομηνίε. Αυτά. Ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία τους και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Well, και προσβλέπουμε στην τελική μορφή της εκθεσής σας. Είπατε 30 Μαΐου είναι η προθεσμία. Ναι, 22 ε, Μαΐου περιμένουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το έχουμε και αυτό υπόψη, γιατί μπορεί να μας δώσει κάποιες ιδέες η ανακοίνωση της Επιτροπής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση και πάμε στο επόμενο σημείο που έτσι πάρα πολύ εύκολα θα πάρω το ρόλο του εισηγητή τώρα. Στο σημείο 6 στήσουμε τις τροπολογίες για τη γνωμοδότησή μου σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας και επικαιροποίηση οδηγία γιατί κάποιον τους κανονισμούς που διέπουν τα σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη. Είναι όλοι παρόντες εδώ, οι σκιώδεις και όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Έχουμε και τον εκπρόσωπο της ΓΔ επιχειρήσεις, ο κύριος Ζηράου είναι ο επικεφαλής. Βλέπω και τους ειδικού επί του θέματος που θα πάρουν το λόγο σε λίγο. Να ξεκινήσω εγώ τη συζήτηση σχολιάζοντας τις τροπολογίες. Δεν ε, θα πω και πάλι τα γενικά σχόλια που έκανα όταν παρουσίασα τη γνωμοδότηση, μάλλον θα πρέπει να εστιάσω στις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα, από τις 66 τροπολογίες, ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών είναι δική μου πρωτοβουλία, όμως ευχαριστώ πολύ και άλλους συναδέλφους και τους σκιώδεις που προσεπέγραψαν πολλές από τις τροπολογίες μου. Εργαστήκαμε πολύ στενά με τους σκιώδεις για να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση από κοινού. Οι δικές μου τροπολογίες αφορούν κατά κύριο λόγο την εισαγωγή ε, των ε, ιδεών για ε, τις νέες κατηγορίες σχεδιασμού και είχα με πολύ θετική ανταπόκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε οι κατηγορίες σχεδιασμού να είναι πιο ξεκάθαρες και να συνδέονται, αν θέλετε καλύτερα, με τις συνθήκες που πρόκειται να εκπληρώσουν τα σκάφη αναψυχής. Κυρία αν θέλετε, μας υπέβαλε μια ελαφρά διαφορετική τροπολογία επί του θέματος. Για τα ποντοπόρα σκάφη και πιστεύω ότι είναι πολύ συγκεκριμένη η άποψή μα σχετικά με τις προϋποθέσεις που αφορούν τον άνεμο. Σχετικά με τον άνεμο και το ύψο των κυμάτων, διότι ε, υπάρχουν συνθήκες ε, βάσει των οποίων μπορούν να κατασκευαστούν τα σκάφη είτε για βαθιά είτε για ρηχά νερά. Βεβαίω θα περιμένουμε να δούμε τι, ποια είναι η γνώμη του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Υπάρχουν και ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με τη σήμανση και άλλες, άλλα θέματα τα οποία έχω συμπεριλάβει και δεν χρειάζεται να σχολιάσω αλλά όποιος θελήσει να θέσει ερωτήσεις είναι φρόσδεκτος. Θέλω τώρα να επισημάνω ορισμένες άλλες τροπολογίες που έχουν προτείνει οι συνάδελφοι. Ο κύριος Μάντερς έχει υπάρξει ο πιο δραστήριο στο θέμα των τροπολογιών και θέλω να του πω ότι ενώ συμφωνώ με την ιδέα του, της, ε, της εναρμονισμένης αδειοδότησης ε, για την ε, ναυσιπλοεία νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιληφθεί ε, την εισαγωγή και τα εκτιμώντας και μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο άλλο σημείο η μνή αυτή. Επίσης μιλάτε για θέματα φοροδιαφυγής για τον ντίζελ και δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με την πρόταση αυτή αλλά θα επανέλθω στο σημείο αυτό αργότερα. Υπήρχε και μία τροπολογία σχετικά με τις ευθύνες σχετικά με την σήμανση της γραμμής πλεύσεως και ε, δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να ζητήσουμε ευθύνες από τον κατασκευαστή. Ο κύριος Σβάμπ έκανε ορισμένες προτάσεις για την, ε, τον εντοπισμό των ε, σημείων της χώρας προελεύσεως και ε, των πιδενακίδων κυκλοφορίας και τέλος ο κύριος Σβάμπ έχει κάνει κι άλλη μία, μία τροπολογία σχετικά με τον μηχανισμό ε, ε, επιγούσης στάσεως και ε, νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί γενικά στα θέματα αυτά και δεν χρειάζεται να περιληφθούν. Αναφέρθηκα λοιπόν στις τροπολογίες, πιστεύω όμως ότι γενικώ τώρα έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία με ευρία συνένεση και μετά θα συζητήσουμε την Επιτροπή πώς θα προχωρήσουμε προχωρήσουμε διότι ε, θα ψηφίσουμε στην Δανική Προεδρία. Δεν μας έχει ενημερώσει η Κυπριακή Προεδρία για την πρόοδο του θέματος στον τομέα τους και πρέπει να δούμε αν ακολουθούν την ίδια πορεία που ακολουθούμε και εμείς. Ίσως σας ενδιαφέρει ότι τη Δευτέρα που ήμουνα στην Κοπενχάγη συνάντησα την ε, Δανέζα ε, Υπουργό Περιβάλλοντος για τον θόρυβο και τα καυσαέρια και αυτά ε, τα θέματα ήθελα να θίξω κατά την παρουσίασή μου και τώρα καλό τους και όδους εισηγητές ε, να επέμβουν ξεκινώντας από τον κύριο Σουάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, νομίζω ότι ήδη έχετε επισημάνει τις βασικές τροπολογίες και νομίζω ότι η τροπολογία 52 για σκάφη τα οποία αθλητικά σκάφη που μπορούν να κινηθούν μόνο στη χώρα κατασκευής τους ε, δεν είναι φιλική προς τον καταναλωτή. Επίσης όσον αφορά αυτή την επίγουσα δυνατότητα στάσεως ε, είναι μια ρύθμιση η οποία θεωρώ ότι ε, είναι σκόπιμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον ήθελα να αναφερθώ στην εισαγωγή των νέων κατηγοριών 59, 61, 62 και 63 και στις τροπολογίες αυτές βλέπουμε ότι ε, θα πρέπει να φροντίσουμε σχέτως του briefing το οποίο ζητούμε θα υπάρξει ψήφιση των ε, τροπολογιών. Εάν δεν είναι ε, σκόπιμη η θέσπιση αυτών των μέτρων προτείνω τροπολογία 56, ιδίω για τα υβριδικά μέσα κίνηση και καύσιμα και αυτά είχα να πω μόνο κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ κύριο Δρέπο. Θα ήθελα... Ήτανε μία πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε κάποιον εμπειρογνώμονα να τοποθετείτε για αυτό το ζήτημα. Η κυρία Κορχόλα και ο υποφαινόμενος καταθέσαμε σχετική ε, τροπολογία από πλευράς ε, των ε, ε, κομμάτων ε, στην Φινλανδία που επιθυμούσαν μεγαλύτερη ασφάλεια για τα σκάφη αναψυχής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εναλλακτικέ λύσεις για την αναβάθμιση της ασφάλειας ε, μας βρίσκουν σύμφωνους. Γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα για την προσαρμογή της, προς αυτή την κατεύθυνση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα προσέθετα ότι όλα είναι συνάρτηση του θαλασσίου χώρου και επίσης των καυσίμων που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια μιλάμε για την μείωση των ε, εκπομπών αερίου την επόμενη πενταετία. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, όλα ε, στην ουσία τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως σας έλεγα, μας βρίσκουν σύμφωνο Σε παραδείγματο χάρη ε, ηλεκτρική, ένα ηλεκτρικό κύκλωμα για την ασφαλή πάυση λειτουργίας του κινητήρα, Πιστεύω ότι όλα αυτά τα μέτρα θα είναι προς όφελος ε, και των κατασκευαστών. Στη Φινλανδία ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές κατασκευαστικές εταιρείες και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάνδρης τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που νομίζω ότι είμαι σκιώδης. Ε, όταν είναι κάποιο δραστήριο, όλοι νομίζουν ότι είναι ή συγητή ή σκιώδη. Χαίρομαι λοιπόν που θεωρείτε ότι είμαι δραστήριο. Ε, δεν είναι πολύ αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Ε, ζήτησα κάποια πράγματα για να προσθεθούν μέσα στα εκτιμώντας ε, μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειε όταν έχουμε ολοκληρωμένε προτάσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλάμε για τυποποίηση και ενίσχυση τη ασφάλεια κτλ., ξεχνάμε το πιο σημαντικό, του ανθρώπου που χρησιμοποιούν τα σκάφη ή τα ποδήλατα ή οτιδήποτε. Ε, θα μου πει κάποιο ότι δεν είναι η εντολή μα. Αλλά δεν μπορούμε να ε, ξεχνούμε τους ε, χρήστες, παρότι αυτό όντω δεν ε, εμπίπτει στην εντολή μας. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να εισηγηθεί λύσεις. Εσείς που είστε οι εισηγητής, νομίζω, ελπίζω τουλάχιστον, θα υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου. Είναι μια ισοσκελισμένη πρόταση και Χαίρομαι. Ο κύριος Χάρμπορ. Δεν είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ευθύνη των κρατών μελών ε, να διεξαγάγουν συστηματικού ελέγχου, να διοδοτούν, ε, να ε, εκπονούν τεχνικέ προδιαγραφέ. Τέλο πάντων, θα τα πούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Ρούλε. Λοιπόν, εγώ Θέλω να απαντήσω εδώ στον κύριο Μάντερς. Έχω πρόβλημα με την τροπολογία 58, διότι πρόκειται για ένα άρθρο και όχι για τα εκτιμώντας και θα ήθελα να ξέρω πώς αυτό μπορεί να μεταφερθεί στα εκτιμώντας. Δηλαδή, εφόσον νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των διπλωμάτων οδηγήσεως πλεύσεως θα πρέπει να δούμε τι μελγενέστε στηρίζουμε και άλλες ε, ε, ε, και άλλα θέματα αλλά θα περιμένουμε το briefing paper προτού εκφραστούμε επί του θέματος αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ Ευχαριστώ. Και εγώ ξέχασα να μιλήσω για το briefing paper, το οποίο επίκειται. Θα δούμε πώς αυτό προβλέπετε. 30 Μαΐου είπατε. 30 Απριλίου, ωραία. Λοιπόν, το briefing paper θα είναι έτοιμο στον ούπο, την επόμενη εβδομάδα οπότε θα το κοινοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να δούμε αν υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη στις συμβιβαστικές τροπολογίες συμπεριλαμβανομένων των σχολείων του κυρίου Λέμπο και της κυρίας Κόχολα βέβαια θα ενημερώσουμε δεόντως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλα σχόλια τότε ο κύριος Ζεράρ έχει το λόγο για να σχολιάσει την πρόταση αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο από το Συμβούλιο εδώ, αλλά ίσως θα θέλατε να μας πείτε τι γίνεται στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου επί του θέματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία ε, για να κάνουμε σχόλια Οπότε ε, θα κοιτάξω τις τροπολογίες, θα σας ενημερώσω και για το Συμβούλιο όπου πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της ανάλυσης σχετικά με τα άρθρα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στα παραρτήματα. Οπότε πιστεύουμε ότι μία ή δύο συνεδριάσεις στο πολύ της ομάδος εργασίας θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση της οδηγίας αυτής και των παρατημάτων αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ως προς τις συνεδριάσεις που θα θελήσει να οργανώσει η επόμενη Προεδρία. Πιστεύουμε ότι η πρώτη συνεδρίαση θα μπορέσει να διεξαχθεί το Σεπτέμβριο και θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τη νέα Προεδρία να οργανώσουμε την εργασία κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό πριν τελειώσει το έτος. Όσον αφορά τις τροπολογίες, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένες που μας προβληματίζουν περισσότερα. Καταρχήν είναι οι τροπολογίες 41 και 48, δηλαδή το θέμα των κατασκευαστών και πρόκειται για θέματα εφαρμογής και διαπιστώνουμε τώρα ότι αναπτύσσουμε στα εκτιμώντας ένα θέμα που αναφέρεται και στα άρθρα και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ερμηνείας και να ερμηνευθεί κατά τέτοιο τρόπο όπου θα λέγεται ότι όλα όλες οι κατασκευαζόμενες μηχανές για θαλάσσια χρήση ε, θα πρέπει να ε, ελέγχονται για να δούμε το ύψος των καυσαερίων και ενδέχεται να λεχθεί ότι ε, αυτά λέει ο κατασκευαστής εδώ αλλά εμείς πρέπει να τα ελέγξουμε για να δούμε ότι δεν υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί. Οι δοκιμές αυτές είναι δαπανηρές και θα είναι πρόβλημα για τους μικρούς κατασκευαστές. Γι' αυτό και θα προτιμούσαμε το θέμα αυτό να παραμείνει στις εφαρμοστικές διατάξεις, να μην είναι ε, να χρειάζεται απλώς να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο όπου θα καθορίζονται ποιες μηχανές πρέπει να ξαναεξεταστούν και που δεν χρειάζεται άλλη τέτοια εξέταση διότι όπως σας είπα οι δοκιμές αυτές είναι δαπανηρές. Το θέμα των αδειών όπως σας είπα αυτό είναι και των διπλωμάτων είναι ε, θέμα των αρχών μεταφορών δεν θα συζητήσουμε εδώ το θέμα γιατί δεν εμπίπτει στην εμβέλεια αυτής της οδηγίας όσον αφορά τις ε, τροπολογίες 64 χώρα κατασκευής θέλουμε να διατηρήσουμε το κείμενό μας διότι πέραν των ε, άλλων ε, επιχειρημάτων οι ε, ε, αρχές που εποπτεύουν την αγορά θα θελήσουν ενδεχομένως να επισκεφτούν τον κατασκευαστή και η χώρα του κατασκευαστή είναι σημαντική στο θέμα αυτό. Μετά όταν μιλάμε για εξολέμβια που οδηγούνται και θα πρέπει να υπάρχει ένα μέσο να σταματήσει κανείς ε, τη λειτουργία της μηχανής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιομορφίες αυτών των μηχανισμών που σταματούν ε, την κίνηση και ε, όσον αφορά τις τροπολογίες 48 και 51 ε, μάλλον 43 και 51 ε, τονίζουν θέματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επιληθούν εδώ γιατί το θέμα της σημάνσεως συζητείται σε ένα από τα εκτιμώντας όπου μιλάμε για τις, ε, τη σήμανση της γραμμής πλεύσεως που είναι θέμα του κατασκευαστή και δεν είναι θέμα της ε, εποπτείας ε, της αγοράς όπως λέγεται στην τροπολογία 43 για το 51 όσον αναφορά αφορά τις επιθεωρήσεις. Είναι θέμα της αρχής εποπτείας της αγοράς και μπορούν ανα πάσα στιγμή οι αρχές αυτές να επέμβουν. Είναι στην διακριτική τους ευχέρεια να επιθεωρήσουν. Όσον αφορά τις δοκιμές κατά την αγορά, τροπολογίες 53 και 58, θεωρούμε ότι είναι περιτές διότι όταν ε, όταν και αν χρησιμοποιηθούν βιολογικά καύσιμα ή στην αγορά τότε θα χρειαστεί να εκπονήσουμε και δοκιμές για να προσαρμόσουμε σχετικά την νομοθεσία. Όσον αφορά την τροπολογία 56 συμφωνούμε. Θα θέλαμε απλώς να προτείνουμε μία διατύπωση σχετικά με ε, τα αποτελέσματα. υπάρχει ένα σύστημα για την, τον σχεδιασμό των σκαφών και θα πρέπει αυτό να αντικατασταθεί με κάτι άλλο άπαξ και έχουμε την σχετική έκθεση. Ε, τροπολογία 57. Η καθυστέρηση την οποία προτείνουμε είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προτείνει η έκθεση και πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις ε, μέσες τιμές ε, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Εάν μου επιτρέπετε όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην τροπολογία 32 διότι συμφωνούμε με τους στόχους ότι δηλαδή θέλουμε να αναφέρουμε το κίνδυνο παλινδρομήσεως και αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευκρινίζει ότι χρειάζεται είτε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παλινδρόμησης και ε, στην αντίθετη ε, περίπτωση να δούμε εάν το σκάφος έχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να μπορέσει να παραμείνει ε, εν πλώ και να μην βυθιστεί. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ο κατασκευαστής να πάσα στιγμή πρέπει να προβεί σε μία ανάλυση του κινδύνου και να αποδείξει είτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ή αν υπάρχει κίνδυνος έχουν, έχουμε εξασφαλίσει ότι αρκεί η δυνατότητα διατηρήσεως του πλοίου ε, του σκάφους ε, εν πλώ. Και δεν έχουμε αντιρρήσεις στις άλλες τροπολογίες, απλούστατα θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Άλλα προβλήματα δεν έχουμε. Αν όμως μου το επιτρέψετε, θέλω να κάνω μία αναφορά σχετικά με το γεγονός ότι μιλάμε ε, για πόντοπόρα και άλλα. Φόσον λοιπόν οι ενδιαφερόμενες κοινωνικές τάξεις το θεώρησαν απαραίτητο, πιστεύουμε ότι στην τροπολογία 44 η αναφορά ε, ότι οι χαρακτηριστισμοί αυτοί μπορεί να δημιουργήσουν παρανοήσεις είναι περιττός, διότι είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τους ενδιαφερόμενους. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και περαιτέρω εάν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, πραγματικά εξελικτική απάντηση για όλες τις τροπολογίες. Οπότε να βγάλω κάποια συμπεράσματα με τους συναδελφούς. Κύριε Αστράου και Μάντερς, μπορείτε να με έχω την προσοχή σας μια στιγμή ως σκιώδης σύγητες. Πρώτα απ' όλα, ακούστηκε μια σημαντική πληροφορία από την Κομισιόν ότι εξειδικευμένες μα εργασίες έχουν επιτύχει μια κάποια πρόοδο. Οπότε κύρια, η επόμενη κύρια συνεδρίαση θα γίνει το Σεπτέμβρη, άρα έχουμε μια κάποια εικόνα για το χρονοδιάγραμμα. Έχω την αίσθηση ότι δύο είναι οι παράγοντες που με κάνουν να προτείνω να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή για κάποιες εβδομάδες. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση αξιολόγησης δεν θα την έχουμε πριν τις 30 Απριλίου. Και δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο ουσιαστικά για να την μελετήσουμε έως 30 Μαΐου. Επίσης θα θέλαμε να δούμε τις γνωμοδοτήσεις ε, των Επιτροπών Μεταφορών και Περιβάλλοντος που ψηφίζονται σήμερα ή αύριο. Και η ομάδα εργασίας πιστεύω ότι πρέπει να ξαναεξετάσει κάποιες τροπολογίες. Καλό λοιπόν είναι το Σεπτέμβρη Καλό είναι η ομάδα εργασία να μπορέσει να έχει χρόνο να ξαναδεί κάποια ζητήματα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να περάσουμε αυτό το κείμενο στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε και με την Κυπριακή Προεδρία. Οπότε εγώ προτείνω αναβολή, αν συμφωνούν και οι σκιώδεις, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πλήρως όλες τις πτυχές της έκθεσης και να ζητήσουμε και κοινή συζήτηση και με τους ενδιαφερόμενους από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Και με χαρά να προσκαλέσουμε και την Κομισιόν να συζητήσουμε τα θέματα και εκείνη τη στιγμή. Γιατί από ό,τι μας είπε, ήδη είχε μια σαφή τοποθέτηση για συγκεκριμένες τροπολογίες. Ελπίζω να καταλήξουμε στο τέλος σε ευρία συνένεση του εγγράφου και θα μας ενημερώνει βεβαίω και για τις εξελίξεις στην ομάδα Συμβουλίου. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα σας αποστείλω αγαπητοί συνάδελφοι ένα νέο χρονοδιάγραμμα, ώστε οι να έχουν αρκετό χρόνο να μελετήσουν όλα τα θέματα αυτά λεπτομέρω. Μια μισή με δύο ώρες ε, συνεδρίαση σκιωδών. Αν ε, δεν υπάρχει διαφωνία, αυτό θα κάνουμε λείπει, οι υπόλοιποι σκιώδεις είναι εδώ και συμφωνούν. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις πληροφορίες. Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε ουσιαστική πρόοδο σε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Λοιπόν, είμαστε πέντε λεπτά πριν το χρονοδιάγραμμα, όμως η κυρία Μακλάρκιν είναι εδώ, είναι η συγγήτρια για το ΣΥΒΕΦΤΑ. Να ξεκινήσουμε λιγάκι νωρίτερα. κύριος Ρέπο, κύριος Μπαλτασάρη, κύριος Σμιτ όχι, κύριος Μάντρες θα μείνει, κύριε Σερούτα και ο κύριος Σμιτ είναι εδώ. Sorry, yes, you slipped in. Μπήκατε και δεν σας κατάλαβα. Γιατί σας έψαχνα και νωρίτερα. Mm. Είσαστε ο προσκεκλημένος κοιόδης σήμερα. Λοιπόν, οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε αν είναι ήδη παρόντας. ποιον περιμένουμε. Mr. Mr. Herbert. Τον κύριο Herbert. Mr. Herbert is here. Okay. Oh, yes, sorry, sorry. Yes, I saw you there. Yes, okay. Well, so the full cast is assembled. So... Είναι άπαντες παρόντες, οπότε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μακλάρκεν να μας παρουσιάσει τη νέα γνωμοδότηση για το πρόγραμμα για την αγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2020. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ανέλαβα αυτή τη γνωμοδότηση που έχει αντικείμενο την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με καλύτερη ε, πρόσβαση στην χρηματοδότηση ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα ιδίω στι ομάδε στόχου που είναι οι νέοι και οι γυναίκε και να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και παγκοσμίω. Αυτό είναι ένα άλλο από του στόχου που υποστηρίζω στο τομέα αυτό. Είναι σαφέ ότι η ε, αυτοπασχόληση και η επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασία. Παρά τα αυτά, σε τέτοιου χαλεπού περισσότερη ανάπτυξη, αλλά και καλύτερου όρου για την επιχειρηματικότητα, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και του ε, πολίτε που θέλουν να δημιουργήσουν δική του επιχείρηση. Εγώ θα ήθελα η γνωμοδότηση αυτή να εστιάσει παρά τα αυτά σε πολύ συγκεκριμένου τομεί, για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό κλίμα επιχειρηματικότητα θα ήθελα εγώ να εστιάσω ιδίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, που πολύ συχνά λέμε ότι είναι η ραχοκαλιά τη ευρωπαϊκή οικονομία. Στην πρόταση αυτή πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό με πολλού τρόπου που θα σα παρουσιάσω τώρα. Μπορούμε να προωθήσουμε επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όχι μόνο στην ανακτήριό του φάση, αλλά όχι μόνο στην φάση ανάπτυξη, αλλά και στην ανακτήριο φάση, στο startup όπου το κόστος της ίδιας της επιχείρησης είναι πάρα πολύ ψηλό. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν προσπαθεί ε, να ε, κάνει σχετικές προτάσεις, αλλά μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές με το ξέρω των μελών για να δούμε καλύτερα πώς γίνεται η κίνηση επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα. Έπειτα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις ενημερώσουμε καλύτερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να βοηθήσει για να εντοπιστούν τρόποι χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξη ταγωνιστικότητα. Περισσότερη καθοδήγηση μπορεί να δοθεί επίσης για πολλά ζητήματα όπως ε, φραγμή στην είσοδο στην αγορά, θέματα προτύπων, ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Να, να, να τα λέω πιο αργά. Τι ωραία, έχω όλη τη μέρα άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις εν γέννη. Πάντως δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη μέτρων, μέτρων δηλαδή που ήδη έχουν θεσπίσει τα κράτη-μέλη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα αποτελέσματα της άσκησης χαρτογράφησης που κάνει η Κομισιόν ώστε να ελέγξουμε ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή ώστε αυτό το πρόγραμμα να έρθει να λειτουργήσει ως προστιθέμενη αξία. Τώρα, για τα μέτρα απλούστευσης. Θεωρώ ότι η έξυπνη νομοθεσία και τα fitness checks είναι πάρα πολύ σημαντικά. σαν αντικτύπου για τα ενωσιακά μέτρα και να δούμε πώς επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Άρα, να δούμε πώς μπορούμε να καταργήσουμε και την νομοθεσία και να πλουσιάσουμε νομοθεσία ώστε να αρχιστοποιηθεί το άχθος εκεί όπου είναι αναγκαίο. Έπειτα, ε, ειδικέ δοκιμές που να μπορούμε να μετρούμε με αυτές την ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πάρα πολύ σημαντικές δηλαδή δυνατότητες για να μειωθεί το σχετικό άχθος. Το One Stop Shop που ήταν μια παλιά πρόταση Κομισιόν ε, είναι κάτι που με απασχολεί. Θέλω όμως να ακούσω πιο πολλές ε, διευκρινήσεις και από την Κομισιόν και από τους σκιώδεις σχετικά με το κόστος. Δεν θα ήθελα να έχουμε επικαλύψεις, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσει σε εφιστάμενα ε, website που υπάρχουν στα κρατημέλη και όχι να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν κάτι άλλο. Πώς θα αντιμετωπίσει στατιστικά στοιχεία που εντόπισα ότι στις ΗΠΑ έχουμε πενταπλάσιες επενδύσεις σε κεφάλαια κινδύνου σε σχέση με ότι επενδύουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν προκειμένου για να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω για τον τουρισμό. Είμαι αρκετά ε, διστακτική εν προκειμένου και οι Σκιώδης ε, και η Αρμόδια Επιτροπή α, διαφωνούν, καθώς υπάρχουν πολλές, πολλοί κλάδοι, πολύ πιο σημαντικοί εν προκειμένου που δεν αναφέρονται. Έπειτα θα υποβάλω τροπολογίες για τον αντίκτυπο για την ανάπτυξη και τις θέσει εργασία ε, και για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα το πώς οι στόχοι του προγράμματο έχουν επιτευχθεί. Θα αποστείλω προς μετάφραση το κείμενό μου την πέμπτο απόγευμα. Είναι σχεδόν λοιπόν ε, τελειωμένο το κείμενό μου, αλλά θέλω να ακούσω πρώτα απ' όλα τις θέσεις των σκιωδών σε σχέση με όσο είπα σήμερα και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θέλουν να θέσουν ως προτεραιότητα στις τροπολογίες. Παρακαλώ λοιπόν να μου στείλετε έως αύριο τις ε, προτάσεις σας, ώστε να τα λάβω υπόψη πριν αποστείλω το κείμενό μου στη μετάφραση θέλω πραγματικά να ακούσω τι δικέ απόψει. Τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα, ώστε να μπορέσουμε οι επιχειρήσει και οι δύο μικρομεσαίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμείνουν ανταγωνιστικέ. Ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed, Mrs. McClarkin. Κυρία Μακλάρκιν, ε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία και είχατε ήδη και κάποιε ιδέε για να συζητήσουμε επιμέρου τροπολογίε. Για να ακούσουμε τώρα του ε, σκιώδει. Ο κύριο Μπαλτεσάρη θα αρχίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά η πρόταση αυτή για την συνέχιση του προγράμματος COSME ακολουθώντας αυτά που έχουμε ήδη θεσπίσει είναι πραγματικά κάτι που ε, θέλω να επενέσω. Το πρόγραμμα Κόσμο ουσιαστικά βασίζεται στα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και θέλει να βελτιώσει την... Ε, τα ελλείμματα και, και τα κενά. Είναι ένα πρόγραμμα αυτό το οποίο στοχεύει πιο πολύ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια οικονομικής κρίσης όπου το πρόβλημα ε, της εξέβρεσης χρηματοδότησης είναι γενικευμένο με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Οπότε το πρόβλημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τους επενδύσεις του και την γενικότερη δραστηριότητα είναι κάτι θεμελιώδους σημασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να προβλέψουμε και άλλα μέτρα που να συνδέουν τα εργαλεία που προβλέπει αυτό το πρόγραμμα με τα εργαλεία που ήδη διαθέτουν τα κράτη-μέλη, όπως είναι τα εργαλεία συνοχής ή άλλα εργαλεία εθνικής πολιτικής. Τι θα μπορούσα να πω. Ένα δις και 400 εκατομμύρια ε, πάνω από τα 2,5 δις υπέρ των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα εύλογο ποσόν αλλά θα έπρεπε να είναι περισσότερο θεωρώ. Μια από τις βασικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η παρακολούθηση ε, της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων. Αυτή η κατανομή λοιπόν, ε, η σωστή κατανομή θα μπορούσε να είναι ένας από τους στόχους τη δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, θεμελιώδου σημασία είναι να συνδέσουμε σε όλα αυτά και την διοικητική απλούστευση που ακόμη και τώρα καθιστά τη δημιουργία επιχειρήσεων πολύ χρονοβόρα και ε, θέτει επίσης πολλά περιτά βάρη ε, που ε, δημιουργούν εμπόδια στην άμεση χρηματοδότηση. Θεωρώ επίσης ότι καλό είναι να αναφερθεί και ο τουρισμός μεταξύ των τομέων τους οποίους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Γι' αυτό το λέω. Δείτε ποιο είναι το ΑΕ που παράγει ο τουρισμός. Ιδίω σε σχέση με τις νέες ε, αρμοδιότητες που απορρέουν για την Κομισιόν από τη νέα Συνήθιση Λισαβόνας. Δείτε το αυτό. Μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε μεγαλύτερη προσοχή αυτό το ζήτημα. Μην βλέπετε τα πράγματα υπό το μικροσκόπιο των συμφερόντων της δικής σας χώρας, αλλά υπό το, υπό το πρίσμα του γενικότερου ευρωπαϊκού συμφέροντος. Έπειτα, πολύ εύλογο θα έλεγα ότι είναι και ο στόχος ε, που λέει ότι μέσω συγκεκριμένων φορέων όπως εκείνοι που δημιουργήθηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα θα μπορεί να δοθεί μια όθηση στην εξωτερήκευση και στην εξωτερική δραστηριότητα των ε, επιχειρήσεων ώστε να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην ε, δημιουργούμε εμπόδια, εμπόδια συγγνώμη, ε, που δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το ψηφιακό μέρισμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι και ευκαιρία. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε μόνο θύματα της παγκοσμιοποίησης. Είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και μπορεί να επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βγουν από το επαρχιακό τους καβούκι και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πλήρως α, αυτές τις δυνατότητες τέτοια δίκτυα, όπως το δίκτυο για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρξει και ένα εργαλείο στήριξης για τη δημιουργία δικτύων ή συμπράξεων, κοινοπραξιών μάλλον, μικρών επιχειρήσεων, ώστε να καλυφθούν, να γεφυρωθούν ή ε, τα χάσματα που υπάρχουν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μια μικρομεσαία επιχειρήση για να διεισδύσει σε αλλοδαπές αγορές. Πώς μια μικρομεσαία επιχείρηση από μόνη της να ε, διεισδύσει στην κινέζικη ή σε λοιπές ασιατικές αγορές. Μόνο με μια τέτοια υποστήριξη. Βεβαίως, εξίσου σημαντικός είναι και ο σκοπός αυτού του προγράμματος που αφορά την προώθηση της ε, αυτοαπασχόλησης και πώς συνδέεται αυτή με την επιχειρηματικότητα, άρα να αρθούν τα περιτά γραφειοκρατικά εμπόδια, ειδικά σε ένα περιβάλλον κρίσης που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες νέα επιχειρηματικότητας. Ήτρια έμφαση θέλω να δώσω στην παρακολούθηση και την επαλήθευση. Στο παρελθόν, η επαλήθευση ε, κατέδειξε τη σημασία και τη λειτουργικότητα ενός προγράμματος. Και εδώ επανέρχομαι πάλι στο θέμα της χρηματοδότησης και της προώθησης των επιχειρήσεων. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Δρέποτα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κρίνω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων μέτρων. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι βάσει των τελευταίων ε, μελετών 2002-2010 προκύπτει ότι περίπου 25% των νέων θέσεων απασχόλησης δημιουργήθηκαν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Φινλανδία. Το αντίστοιχο ποσοστό ε, ανέρχεται στα 90%. Οι μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις είναι ο πραγματικός ε, κινητήρας της μελλοντική ανάπτυξης. Από στρατηγικής πλευράς ε, είναι απαραίτητη εταίρη για μας ε, ε, με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής 2020. Προετοιμάζεται τώρα αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω όμως ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των περιορισμένων πόρων. Γιατί δεν θα διοχετευθούν οι πόροι μόνο σε αυτούς που εξασφαλίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη και που ε, χρησιμοποιούν την τεχνολογία εχμής, δηλαδή οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται ήδη σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να διεσυνδεθεί με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 διότι οι πόροι είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με το πρόγραμμα που τώρα προετοιμάζουμε. Καταλαβαίνω ότι με μεσούσεις ε, της κρίσης ε, δύσκολα μπορούμε να ε, επιδιώξουμε αύξηση των πόρων για το πρόγραμμα COSME, αλλά Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια, το κονδύλι δηλαδή που έχει προβλεφθεί για ολόκληρη ε, την περίοδο προγραμματισμού είναι πολύ χαμηλό, κυρίως όταν το αντιπαραβάλλουμε με ε, τα 80 ε, δισεκατομμύρια του προγράμματος ε, ε, και τα 2 δισεκατομμύρια που θα διοχετευτούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν τροποποιηθεί λοιπόν ε, η πρόταση, αν δεν αυξηθεί το κονδύλι, το κόσμο θα είναι ένα εξοραϊστικό και επιφανειακό πρόγραμμα. Δεν θα έχει ουσία. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ε, στην ε, συνέχεια, όταν προχωρήσει η εξέταση του πράγματος, ε, θα τοποθετηθούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και χάρη στη δουλειά της κυρίας Μακλάρκιν ελπίζουμε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα που θα μας βοηθήσει πραγματικά να υλοποιήσουμε τη στρατηγική 2020. Ευχαριστούμε κύριε Ρέπο, κύριο Σμιτ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ορισμένες φορές θεωρώ ότι μιλάμε υπερβολικά αλλά δεν κάνουμε αρκετά. Πιο πολύ μιλάμε παρά ενεργούμε και αυτό που κάνουμε με τις προτάσεις δεν, δεν μεταφέρεται σε αυτούς που χρειάζονται τις προτάσεις και τις αλλαγές και αυτό είναι το πρόβλημα. Πέρυσι Ήμουν επικεφαλής και πρόεδρος ενός σεμιναρίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί υπήρχαν ε, οι επιχειρηματίες που είχαν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα αλλά δεν το γνώριζαν. Όλα αυτά βέβαια είναι καλά. και πρόκειται ε, για τη ραχοκοκαλιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως είπαμε. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε εμείς να έχουμε μία πιο θετική αντιμετώπιση και να υπάρξει μία εκστρατεία για συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένους κανόνες και το αναφέρατε διότι ουσιαστικά μιλάμε για μείωση ε, κατά 25% στη γραφειοκρατία για μεγαλύτερη απλοποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επιτύχαμε τους στόχους αυτούς της μειώσεως της γραφειοκρατίας. Είναι κάτι που προωθούμε στη χώρα μου τη Σουηδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ελπίζω ότι η κυβέρνησή μας στην οποία πρόσκυμε το προωθεί αλλά πιστεύω ότι ουσιαστικά ε, δεν είναι εύκολο και ε, πρέπει συγχρόνως ε, να υπάρξει πρόσβαση για τις μικρές επιχειρήσεις στην αγορά, θέματα δηλαδή τα οποία πραγματεύεται αυτή η έκθεση. Το πνεύμα της επιχειρηματικότητας είναι επίσης βασικό, διότι διαβάζω εδώ στο κείμενο ότι μόνο 45% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και λιγότερο από 40% των γυναικών θα ήθελαν να αυτοαπασχολούνται και αυτό το ποσοστό είναι πολύ ψηλότερο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι λένε ότι θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω επικεφαλής σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, να μην είμαι αυτοαπασχολούμενος γιατί τότε θα είναι δύσκολη η ζωή μου και ε, αυτοί είναι οι νέοι, ε, οι ήρωες που δημιουργούν τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και θα πρέπει να τους ανταμείψουμε, να έχουμε ένα ευρωπαϊκό βραβείο σαν ε, συμβολική συνδρομή. Επίσης είχα ακούσει τις απόψεις του κυρίου Ντράγκη, του Προέδρου της ΕΚΤ. Και ξέρετε ότι στην ΕΚΤ έχουν ε, αυτή την διαδικασία μακροπρόθεσμης ανακεφαλαιοποίησης ε, και έχουν ε, κατακριθεί για την έλλειψη ανεξαρτησίας τους. Είπαν όμως ότι τα χρήματα αυτά προβλεπόταν έμεσα να διατεθούν εις την πραγματική οικονομία, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Ελπίζω ότι έχουν βελτιώσει τις προοπτικές. αλλά δεν έχει αυτή η συνδανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, σύμφωνα με τον κύριο Ντράγκη, η κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών σε γενικές γραμμές είναι τόσο κακές ε, ε, και λόγω της προσβάσεως στη χρηματοδότηση. Είναι δηλαδή πολύ επικίνδυνη η πρόσβαση αυτή για να τη χρησιμοποιήσουν. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι πολύ φίλος της κοινή γεωργικής πολιτικής και ε, της πτυχής αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά πιστεύω ότι και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ίσως ο εισηγητής ή η Επιτροπή θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους. Και το επόμενο θα είναι ότι εφόσον είναι επιχειρηματίες θα μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα μέσα που προτείνονται εδώ είναι, αποβλέπουν στη δημιουργία 5.300 θέσεων οργασίες και ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να διευκολύνει τους νέους να καταρτήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε ε, κάτι να μου πείτε επ' αυτού, να μου πείτε κατά πόσον είναι ρεαλιστική αυτή η προοπτική, και αν ε, όντως ε, υπάρχουν ε, αυτές οι 5.300 θέσεις, αν και ο αριθμός είναι πολύ μικρός εν ώψη της ανεργίας που υπάρχει σε ορισμένες χώρες αλλά η ανεργία των νέων είναι το πιο ευαίσθητο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές πολιτικές διαταραχές ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και θα ήθελα τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε. Για τα σχόλια, είπατε ότι εκπροσωπείται εδώ η Κεντρική Τράπεζα από τον κύριο Ντράγκη. Αύριο θα τον δω γιατί ε, ε, μου απίφθηναν πρόσκληση αύριο σε μια σημαντική διάσκεψη στην Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την ε, ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε και υλικό μπορώ να χρησιμοποιήσω αύριο. Η κυρία Πετικάνεν θα προεδρεύει αύριο το πρωί, γιατί θα απουσιάζω όπως σας είπα. Ο κύριος και εγώ είμαι η συγγήτρια, η κυρία Ρούλε ε, και χαίρομαι που θα μιλήσω μετά τον εισηγητή γιατί συμπληρώνω αυτά που είπε. Συμφωνούμε σε πολλά και γενικώ συμφωνώ με την εισηγήτρια. Με ενοχλεί όμως γιατί συνδυάζουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη γραφειοκρατία και έκανα μία μελέτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δικιά μου περιοχή, τη Βάδη Βιρτεμβέργη, για την κατασκευή μηχανών και είδαμε ότι εάν υπάρχει αξιόπεστη πολιτική περιβάλλοντος την σέβονται γιατί τους επιτρέπει να κατακτήσουν νέες αγορές και να προωθηθούν μέσω του ανταγωνισμού. Greening the economy είναι το μήνυμα αλλά θα πρέπει η πολιτική να είναι και αξιόπιστη ε, και συνεκτική και αυτό μου ελέγχθη επανειλημμένος και έρχομαι τώρα ε, στην ε, στην ανεργία των νέων. Εάν τη συνδυάσουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές στα κράτη-μέλη και φοβάμαι ότι μία στρατηγική η οποία παιδίχθη πολύ καλή στη Γερμανία η, κατά της ανεργίας η διητή εκπαίδευση τώρα βάσει της νέας προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάλετε και πιέζεται. Ε, επίσης ε, θα πρέπει όχι μόνο να χρηματοδοτούμε αλλά να εξασφαλίσουμε να έχουμε ε, μία συνεκτική νομοθεσία η οποία να αποτελεί ένα νήμα ενιαίο το οποίο να διατρέχει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε όλους τους τομείς. Όντως υπάρχουν θέματα που έχουν προχωρήσει αλλά αλλά ανέφερθηκα στην αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων ορισμένα θέματα έπρεπε να διερευνηθούν εάν προωθούν ή εμποδίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτό τελείωσα. ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Δίον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να σας χαλάσω την όλη γιορτή που έχετε στήσει εδώ αλλά η θέση μου διαφέρει με αυτή όλων των προλαλισσάντων σε μεγάλο βαθμό ε, και εξεπλάγει διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και με το Εθνικό μου Κόμμα είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά έχω την εντύπωση ορισμένε φορέ ε, ότι οι φιλελεύθεροι έχουν ε, μετατραπεί σε σοσιαλιστέ, οι σοσιαλιστέ γίνονται φιλελεύθεροι, γιατί αν δω τώρα τις αντιδράσεις στη σημερινή συζήτηση, αυτή την εντύπωση αποκομίζω και έχω την... κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα κεντρικό σύστημα σχεδιασμού, αυτό που συζητάμε, ε, που επιτρέπει εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση, ε, καλή απασχόληση για τους δημοσίους υπαλλήλους ε, και θα ήταν κάτι δημοφιλές στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε τι θέλουν ε, οι επιχειρηματίες, δύο πράγματα. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ε, μείωση της ε, γραφειοκρατίας, ούτως ώστε να ξεφορτωθούν όλους αυτούς τους ατελείωτους κανονισμούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που τους δυσκολεύουν και δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, δηλαδή να είναι επιχειρηματίες. Εάν ακολουθήσουμε αυτή την οδό θα κάνουμε αυτό το λάθος. Θέλουμε να υπάρχει καινοτομία, ελεύθερη σκέψη, ε, πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία, ούτω ώστε οι επιχειρηματίε ε, να μετατραπούν σε κινητήρα τη ανάπτυξη. Εμεί εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα, οι γραφειοκράτε και οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την οικονομία και να βοηθήσουμε και τους επιχειρηματίες να εκπληρώσουν το στόχο τους. Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά με την προσέγγιση, διότι αντί να φτιάξουμε άλλο ένα πρόγραμμα, με 2,5 εκατομμύρια ελάχιστο το κονδύλι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. 5.000 ε, θέσει απασχόληση κατά νότα όριο θα δημιουργηθούν ε, με αυτά τα χρήματα και Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ε, καταστήσουμε κεντρική την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, χρησιμοποιώντα ε, ολιγάριθμε ε, πηγέ και αν δεν διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο, δεν θα βοηθήσουμε ε, του επιχειρηματίε. Μιλάτε όλοι για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουμε κινητοποιηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο για να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Μόνο έτσι μπορούμε να τους βοηθήσουμε και κυρίως όχι μέσω ενός τέτοιου προγράμματος φοβούμε ότι αν δεν σημειωθούν ε, ε, αλλαγές ε, θα καταψηφίσω την πρόταση. Σας ευχαριστούμε, ήσασταν ειλικρινέστατος, λέει ο κύριος Χάρμπουρ, τουλάχιστον ζωντανεύετε τη συζήτηση. Ορίστε, σας είδε η κυρία Εύελεν Γκέπχαρτ και σήκωσε το χέρι. Παρακαλώ και στη συνέχεια θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Αφήστε που έχουμε και παρουσίαση. Ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ ότι οι σοσιαλδημοκράτες θέλουν να απελευθερώσουν και θέλω να διευκρινίσω. Είμαστε ε, ούτε για την προγραμματισμένη οικονομία ούτε για την φιλελευθεροποίηση. Βεβαίως πρέπει να φροντίσουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία στο ελάχιστο γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία πλήττει πολλούς πολίτες και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, λύσουμε αυτό το θέμα. Λίγη όμως γραφειοκρατία δεν σημαίνει απορρίθμιση και θα χρειαστούμε κοινού κανόνες. Έχω την εμπειρία συζητήσεων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επισκέπτομαι τακτικά και υπάρχει ένα θέμα που τους ενδιαφέρει πολύ και επαναλαμβάνουν. Ασχέτως των κανόνων αυτό που μας, ενδιαφέρουν, με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει αξιοπιστία, να μην αλλάζουν οι κανόνες κάθε μέρα. να μην αλλάζει από το α στο ω το σύμπαν, να μην αλλάζουμε συνέχεια τις προϋποθέσεις, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να προγραμματίσουμε και να εργαστούμε. Αυτό είναι πολύ πιο βασικό από άλλα θέματα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι βεβαίως Πρέπει να υπάρξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και στον τομέα αυτό βλέπουμε ότι αναπτύσσονται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αγορίες προνομιούχες, niche markets, όπου υπάρχουν, υπάρχει ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα στην κατασκευή μηχανολογικού υλικού που είναι αναγκαία ήδη και χρειάζονται ιδιαίτερη γνώση και εκεί πρέπει να υπάρχει υψηλή ποιότητα. Και το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι όντως ότι η δυνατότητα της χρηματοδοτήσεως στην περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης που διατρέχουμε δημιουργούν πολλά προσκόμματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί είναι ο τομέας στον οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να βοηθήσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε εστιασμένα και συγκεκριμένα να λύσουμε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι πολύ πιο καλύτερο από ότι ένα μεγαλεπίβολο πρόγραμμα το οποίο θα λύσει τα πάντα. Καλύτερα να απαντήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα που τους ενδιαφέρουν πολύ. Σας ευχαριστώ όλους να πω ότι βλέπω με αρκετή κατανόηση το επιχείρημα του κυρίου Γκινιών ότι υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε αυτό το πρόγραμμα και τις γενικότερες πολιτικές μας πρωτοβουλίες για την βελτίωση των ε, συνθήκων πλαίσιο, όπως είναι η πρόσβαση στις αγορές, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πληροφόρηση για τις αγορές υπηρεσιών, απλά σημεία επαφής. Είναι πρωτοβουλίες γενικότερα που χρήζουν, αν θέλετε, άμεσης προώθησης και ενημέρωσης. Επειδή ποτέ δεν μπορώ να αντισταθώ, θέλω και τώρα να σας επισημάνω πόσο σημαντική είναι η χρήση των προμηθειών με τον τρόπο ώστε να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις στις δημόσιες αγορές. Πάντοτε το στοιχείο των δημόσιων αγορών ε, ενέχει και το στοιχείο της επιχειρηματικότητας, θα υπάρχει τροπολογία και ελπίζω να την στηρίξει στη γήτρια. Λοιπόν, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ο κύριο Χέρμπερτ θέλει να σχολιάσει, να πει κανένα δυο λόγια και μετά θα δώσω πάλι και το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω, ε, αν μου επιτρέπετε, σε κάποιε πολύ εύστοχε παρατηρήσει που έγιναν. Πρώτα απ' όλα, ε, εκτιμούμε αυτό που είπατε για το κόσμο, το οποίο έχει έναν μέτριο ε, προπολογισμό, θα έχει το 66% των δράσεων που άμεσα απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση 20% για τις υπηρεσίες προς μικρομεσαίες και το υπόλοιπο που δεν είναι πολλά κονδύλια, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είπατε κύριε Χάρμπερ. Έπειτα, θα ιεραρχήσουμε προτεραιότητες σε τέσσερι τομεί, του οποίου θέλω να φέρω για να απαντήσω στα σχόλιά σα. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ναι, επιχειρηματικό κεφάλαιο κινδύνου είναι ένα από τα διάφορα εργαλεία και το κόσμο είναι ένα από τα πολλά εργαλεία για τη στήριξη των ε, επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου πέρα από τα εργαλεία του ορίου 2020 στα κράτη-μέλη δεν θέλουμε να, έρθουμε, να λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά με τα εθνικά εργαλεία, θέλουμε να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά και να δώσουμε, ε, αν θέλετε, μια διασυνορική διάσταση, λέω στην εισηγήτρια. Δεύτερος στόχος, Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές. Είπατε και εσείς, κυρία Μακλάρκεν, η πρόσβαση στις αγορές είναι πάρα πολύ σημαντική. Η διεθνοποίηση σήμερα, αυτή τη στιγμή, ο κύριος ε, Καγέχα είναι στην ε, Βραζιλία και θα πάει και στη Χιλή. Ε, τον συνοδεύουν εκπρόσωποι 30 επιχειρήσεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνουν οι λατινοαμερικανικές αγορές. Ναι, θα κάνουμε χαρτογράφηση, δεν θα κάνουμε επικαλύψεις. Θα καταστήσουμε διαθέσιμες πληροφορίες. Κάποιοι είπατε και εσεί ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικτυακή πύλη που να ενημερώνει, χωρίς να δημιουργήσουμε μία ε, τερατώδη βάση δεδομένων που θα πρέπει να συντηρείται και τα λοιπά και θα πέτει πόρους. Κύριε Παλτασάρη, ε, για την διεθνοποίηση, πολύ ορθά είπατε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Θέλουμε να εστιάσουμε στη βοήθεια που θα πρέπει να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για, ε, για ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε τέτοιες χώρες. Δεν θα ονοματίσω ποιες είναι οι χώρες αυτές. Άλλη προτεραιότητα, τρίτη κατά σειρά, είναι η της επιχειρηματικότητας. Ένα παράδειγμα του πώς λίγα χρήματα μπορούν να δώσουν μεγάλα αποτελέσματα. Το 2007 μας πήρε 12, χρειαζόταν 12 μέρες για να σταθεί μια επιχείρηση. Σήμερα χρειάζονται 7 ημέρες για τη σύσταση μιας εταιρείας. Κατά μέσο όρο, ναι, ναι, κατά μέσο όρο επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να λανσάρουμε κάποιες δράσεις και να συνεχίσουμε κάποιες άλλες δράσεις από το ΣΥΠ, ε, το Εράσμους. Ε, νέοι επιχειρηματίες χρησιμοποίησαν αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής που φιλοξενούν έμπειροι επιχειρηματίες. Θέλουμε να συνεχίσουμε επίσης το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας ε, να, κάποια παραδείγματα του πώς θα προάγουμε την επιχειρηματικότητα. Τέταρτη προτεραιότητα. Τέταρτη και τελευταία αύξηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα εστιάσουμε σε όλους τους κλάδους, όλες τις μικρομεσαίες, γιατί όλες οι εταιρείε είναι σημαντικές για, για μας. Ε, με αυτό το πρόγραμμα δημιουργούμε και θέσεις εργασίας, ε, κύριε Τεγιόν. Δείκτην έκθεση αξιολόγησης του ΣΥΠ. 170.000 επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΣΥΠ δημιούργησαν θέσεις εργασίας. Κυρία Ρούλε, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Συνεκτικότητα. Η ανταγωνιστικότητα δεν αντίκειται στη βιωσιμότητα. Είναι θέμα συνεκτικότητας όλα αυτά. Συμφωνώ μαζί σας. Τέλος, γιατί ο τουρισμός. Ο τουρισμός ε, διαθέτει ειδικό άρθρο στις συνθήκες Λισαβόνας και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός κλάδος σε πάρα πολλές χώρες μας και θέλουμε και πάλι με λίγα χρήματα ουσιαστικά να ε, προβλέψουμε δράσεις υποστήριξης που θα έρθουν να συμπληρώσουν τις εθνικές δράσεις. Πιστεύω ότι απάντησα ουσιαστικά στα πιο πολλά ερωτήματα. Όμως, με χαρά να δούμε και κάποια θέματα διμερώς, αν ε, θεωρείτε ότι θέλετε να λάβετε και άλλες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σε ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ήταν πολύ χρήσιμη και συνοπτική τοποθέτηση. Θα δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ε, ξέρετε, έχω κατανοήσει για αυτά που λέει ο κύριος Τιγιόν και στο Ηνωμένο Βασίλειο στην εκλογική μου περιφέρεια πολλοί θα ήθελαν να μην μπλεκόμαστε στη ζωή τους, στην καθημερινή τους ζωή, να τους αφήσουμε ήσυχου να κάνουν τη δουλειά τους, να μειώσουν τη γραφειοκρατία, ενώ εμείς φαίνεται ότι την αυξάνουμε. Έχουμε πάντως αυτή την πρόταση και πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε η Επιτροπή Ήτρε Βιομηχανίας να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση τη δική μας, διότι όντως είναι περιορισμένη οι πόροι, είναι 2,5 δις, όχι εκατομμυρία, 2,5 δις. Δεν αληθεύει αυτό που ακούσαμε πριν, δεν είναι εξοραϊστικού χαρακτήρα μόνο το πρόγραμμα, προσπαθούμε να διαχειριστούμε σωστά τα προγράμματα με ανακοινοθέντα τύπου, με διάφορους τρόπους δραστηριοποιούμαστε στον τομέα αυτό. Ε, είναι πολύ επικίνδυνο να ε, διαφοροποιούμε, να ξεχωρίζουμε από όλες τις υπόλοιπες τις βιομηχανίες ε, μία μόνο, γιατί η δράση μας θα πρέπει να είναι οριζόντια και ε, ε, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτό που συζητούσατε εσείς είναι ένα κομμάτι της πίτας, αλλά σίγουρα όχι ολόκληρη πίτα που πρέπει να χωρίσουμε. Ε, Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι να προωθήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα και επανειλημμένα το βασικότερο πρόβλημα είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αφού θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύριο, Μάλκολμ, μπορείς να μεριμνήσεις ώστε να επαληθεύσουν αν ε, δανειοδοτούνται επιχειρήσεις από τις τράπεζες διότι τα χρήματα έχουν χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά για κάποιο λόγο δεν φτάνουν ε, στους αποδέκτες. Ε, σε σχέση τώρα με τον προϋπολογισμό και το κονδύλι. Πιστεύω ότι ε, ο απότερος στόχος θα πρέπει να είναι ε, η απρόσκοπτη πρόσβαση στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μείωση του διοικητικού ε, άχθους, του γραφειοκρατικού άχθους. Πρέπει να ξέρουν όλοι πόσο εύκολα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με ποιο τρόπο μπορούν να την αποκτήσουν. Οπότε με αυτή τη συμβολή ελπίζουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και με αυτό το κονδύλι το 2,5 δις να δημιουργήσουμε όντω περισσότερε θέσει απασχόληση. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Χάρμπορ. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα φύγει για μετάφραση γνωμοδότηση 30-31 Μαΐου ε, θα το επανεξετάσουμε. 7 Ιουνίου είναι η ημερομηνία για τις τροπολογίες ε, και τον Ιούλιο περάσει από την Επιτροπή Ήτρε. Πολύ ωραία. Έχουμε λίγο καθυστερήσει. Ε, θέλω να... Η κυρία Γκάλερ είναι εδώ, σας καλωσορίζω. Δεν έχουμε χρόνο και ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Σμιτ, Σίβιτς... Ε, τέλος πάντων, έχουμε κάποιους σκιώδεις. Ε, μπορούμε... μπορούμε να προχωρήσουμε. Από ό,τι κατάλαβα θα ακούσουμε μια ανακοίνωση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο της πρότασης, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε 20 λεπτά, οπότε προτείνω να εστιαστούμε στην ε, παρουσίαση που θα κάνετε εσείς ε, και θα γίνει μια πληρέστερη ανταλλαγή απόψεων με τους κοιόδης σε επόμενη συνεδρίαση, γιατί δεν ε, υπολείπεται αρκετός χρόνος για να ολοκληρώσουμε. Σήμερα, σε κάθε περίπτωση, θα δούμε. Σας αφήνω τώρα αμέσως να μας παρουσιάσετε την πρότασή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλησα να πάρω το λόγο και μην ανησυχείτε, θα είμαι σύντομη ε, πριν από την παρουσίαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι μπορώ να θέσω ευθύ εξ ε, τα ζητήματα που με ενδιαφέρουν για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το ζητούμενο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει μέσα στον ε, τεχνολογικό αγώνα ταχύτητας ε, που παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα. Η διαδικτυακή οικονομία έχει κέρια σημασία για την απασχόληση πάνω από 800 δις ε, το 2016 ήτι άνω του 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προβλέπουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν μπορεί να παραμείνει θεατή των εξελίξεων λόγω της έλλειψης ρευστότητος ε, στην ενιαία αγορά και έχω κατά νου τις ε, μη ε, διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες ή ε, σε ε, ε, αρκετά φιλόδοξες πολιτικές αποφάσεις. Θα περάσω κατευθείαν στα ουσιώδη. Τέσσερις παρατηρήσεις θα κάνω και στη συνέχεια θα θέσω τέσσερις πρώτες ερωτήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά θα έχει όλο το χρόνο για να τις απαντήσει. Πρώτο θέμα. Ε, καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, χαίρομαι που τα χρηματοδοτικά μέσα της ψηφιακή ατζέντα ε, επιτέλους είναι διαθέσιμα ή μάλλον ε, επιτέλους σχεδιάζονται και ελπίζω να τα καταστήσουμε λειτουργικά ταχύτερο δυνατόν, ώστε τα μελητή να προχωρήσουμε. Μα, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Εγώ ε, επαληθεύω αν λειτουργεί ο τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση. Δεύτερον, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας παρουσιάζει μια κατάσταση όπου σαφέστατα υπάρχει συνένεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει ε, τις ε, πλέον απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές και με τη χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα ε, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στις ε, υποδομές που λείπουν ή που πρέπει να συμπληρώσουμε ούτως ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να λειτουργήσει μόνο εκεί όπου παρατηρούνται ατέλειες και ελλείψεις. Είναι σαφέστατο ότι ο στόχο δεν είναι να επιφέρουμε μεγαλύτερε τρευλώσει στην οικονομία ε, που θα συνιστούσαν και αντικίνητρο για τις επενδύσεις ε, στην ε, αγορά. Επί τρίτον, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο παράρτημα 3 της πρότασης ε, σε αυτό το σημείο η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή μπορεί να προσφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία, διότι στο πρόγραμμα Europeana, όπου υπάρχει πολύγλωση προσφορά υπηρεσιών, λοιπόν, η γενικότητα Δεύτερα, η χρήση των δεδομένων, και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια αγορά 40 δις το χρόνο, ε, είναι ένας τρόπος για να βρούμε ένα αναπτυξιακό μοχλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτο και τελευταίο, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προκρίνει την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και ε, την παρουσιάζει ως κριτήριο για την επιλεξιμότητα των κοινών προγραμμάτων. Θα ακούσω και τους συναδέλφους ε, για όλα αυτά, αλλά θα ήθελα, για να μην καθυστερούμε, να περάσω στις ερωτήσεις που θέλω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτο ακούσουμε την παρουσίαση. Πρώτον, με ποιους ε, εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους μάλλον φορείς έχετε ήδη συναντηθεί. Αυτά τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος ε, που απαριθμούνται στο παράρτημα ε, της ε, πρόταση είναι ένα πρώτο στοιχείο, όμως ε, δεν μας λέτε με ποια κριτήρια κάνατε αυτή την επιλογή. 9,2 δις, ξέρουμε, διοχετεύονται στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με την εξή κατανομή. 7 δις για τα δίκτυα υποδομών και 2,2 δις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωραία. Με ποιο τρόπο αποφάσισε ε, και ε, υλοποίησε αυτή την κατανομή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με στην πρότασή τη ε, εντοπίζει ένα πρόβλημα αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. προσφορά, την προσφορά εύκολα μπορούμε να την ρυθμίσουμε, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της ζήτησης και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει τους καινοτόμους χρήστες να τους προωθήσουμε, ούτως ώστε να επισπευστεί, να μεγεθυνθεί η ζήτηση ε, ψηφιακών υπηρεσιών για να ε, καταστήσουμε τα προγράμματά μας οικονομικά βιώσιμα. Τρίτη ερώτηση, με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εκταμίευση των κονδυλίων από τα κεφάλια, από τα ταμεία. Αν διαπιστώσει ότι στο ίμιση της προγραμματικής περίοδου λιγότερα από τα 9,2 προ να δεις ε, δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί. Ε, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέταρτη και τελευταία ερώτηση ε, μία διαφημιστική εκστρατεία ή ένα επικοινωνιακό σχέδιο έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι νέοι ενδιαφερόμενοι φορείς, γιατί έχω στο μυαλό μου το σωτά ε, θα ήθελα να ακούσω τώρα τις απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως ε, θα ήθελα να λάβω και κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα τέσσερα ερωτήματα. Μακάρι να έχει χρόνο η Επιτροπή να προλάβει και να απαντήσει όλα αυτά τα ερώτημα για να είμαστε δίκαιοι. Κύριε Σμιτ, Ρούλα, Ρούρα, έχετε ερωτήσεις ή σας κάλυψε η κυρία Γκάλο στα βασικά. Ωραία έτσι. Για να είμαι δίκαιος, ρωτώ και τα δικά μου τα σχόλια καλύψατε, αλλά έχω και κάτι άλλο να πω. Το θέμα που τίθεται επιτάπητος είναι πώς θα καλύψουμε το κενό ανάμεσα στις προσδοκίες των κρατών μελών και της Κομισιόν. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το ύψος του ταχύτητα του ευρυζωνικού και κατά πόσον θα το επιτύχουμε, τουλάχιστον θα καταφέρουμε κάτι να επιτύχουμε, να φτάσουμε τα 30 Mbps και τα 100 Mbps τουλάχιστον στα νοικοκυριά κατά 50%. Τουλάχιστον ένα κομμάτι αυτού του φιλόδοξου στόχου, αν μπορούσαμε να επιτύχουμε θα ήταν πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Φίλιππο Μουνιστέρη από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ίνφσο να μας κάνει την παρουσίασή του και να απαντήσει και σε ερωτήσεις. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Σας παρακαλώ να μην ε, ε, όλο το χρόνο σας ε, στις πρώτες διαφάνειες. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι ψήνοπτος και να τα πω απλά, γιατί έχω 15 λεπτά. Και ξεκινάμε πολύ ωραία. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Διευκόλυνση, συνδέοντας την Ευρώπη, ή ΣΕΦ. Άρα, με ρωτήσει κανείς τι είναι το ΣΕΦ, θα έλεγαν πώς θα βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Βλέπουμε έχουμε εντοπίσει μάλλον ένα κενό, όπως το εντοπίζουν κάποιες μελέτες, αλλά είναι 220 με 270 δις είναι το κόστος για να συνδέσουμε ευρυζωνικά όλα τα νοικοκυριά στο 2020. Οι επενδύσεις υπολείπονται, το διαπιστώνουν όλοι. Υπολείπονται σε σχέση με του στόχου. Μόνο 50 δις έως 2020 περιμένουμε να επενδυθούν από τους ιδιώτες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε το ΣΕΦ με συνολικό ε, με 9,2 δις 6 7 για το ευρυζωνικό δίκτυο και 2 3 δις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό θα γίνει με ένα μείγμα επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων. Η επιχορήγηση θα είναι ο βασικός πυρήνας για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ για τις ε, ευζωνικές υποδομές θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα μείγματα επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, ανάλογα με τον τομέα παρέμβασης. Στόχος να μην απομονώσουμε κάτι που δεν μπορεί να δώσει αγορά χωρίς τη δική μας βοήθεια. Γιατί υπάρχουν τομεί όπου δεν είναι οικονομικά βιώσιμοι να παρέμβει μόνο ο ιδιωτικό τομέα. Τα χρηματοδοτικά μέσα θα μα επιτρέπουν να, να ε, κάνουμε μία μόχλευση που υπολογίζουμε για αυτού του είδου τι υποδομέ μπορεί να είναι 6 7 φορέ το ποσό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε 75 εκατομμύρια ε, νοικοκυριά ε, ε, στις ευρωζωνικές υπηρεσίες. Τώρα βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια θα πω λίγα λόγια για αυτές τις επενδύσεις. Γιατί θα κάνουμε επενδύσεις, γιατί το επίπεδο επενδύσεων σήμερα δεν είναι παρκές, δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους νυν παρόχους και τους ανταγωνιστές για τον ενδυνάμει κίνδυνο που ελοχεύει από αυτές τις επενδύσεις και λόγω της οικονομικής ύφεσης που έχει πλήξει πάρα πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Και έπειτα, υπάρχει και ένα πρόβλημα έλλειψης business case στις αγροτικές κοινότητες όπου είναι αεροκατοικημένες και δεν ευνοούν αυτή την επένδυση. Επί τη ψηφιακή υπηρεσία τα πράγματα είναι κάπως πιο ξεκάθαρα. Η Κομισιόν προσπαθεί να δώσει κάποιους, κάποια βασικά στρώματα τέτοιων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Τι ψηφιακέ υπηρεσίε θα τι δείτε στην πρότασή μα στο, βρίσκονται στο ε, νυν πρόγραμμα SIP. Ε, Το SIP αφορά πιο πολύ πιλωτικά project, ενώ από την άλλη μιλούμε για αναπτύξεις μακράς κλίμακας. Βεβαίως κάποιες άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που προτείνουμε είναι εντελώς καινούργιες. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, όπου θα σας διατρέξω σύντομα λίγα στοιχεία για αυτό το χάσμα, αυτό το gap που έχουμε το πίσω ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Αν πάμε να δούμε τι θα συμβεί την επόμενη δεκαετία, θα δούμε ότι δεν γνωρίζουμε τι εφαρμογές θα αναπτύξει η αγορά. Ξέρουμε όμως τι χρησιμοποιεί τώρα η αγορά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τι έχουμε χρηματοδοτήσει μπορεί κανείς να συμπεράνει δικαίως ότι θα χρειαστούν πιο πολλές ευρυζωνικές υπηρεσίες στο μέλλον. Σκεφτείτε, πού ήμασταν πριν από μια δεκαετία. Ποιος θα σκεφτόταν το cloud computing, τα Dropbox ε, στο Facebook και τα λοιπά τέτοιου είδους υπηρεσίες. Είναι ε, συνεχής και ταχύτατη η ανάπτυξη των ε, εφαρμογών και σίγουρα πρέπει να βλέπουμε μπροστά την επόμενη επταετία και πέρα από αυτή. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια και να επισημάνω το εξή. Ήδη υπολοιπόμεθα αρκετά σε ό,τι αφορά το ταχύτατο ευρυζωνικό διαδίκτυο. υπάρχει βεβαίως η ψηφιακή ουδετερότητα γιατί δεν γνωρίζουμε τι είδους τεχνολογία θα χρησιμοποιούμε σε 10 χρόνια. Για παράδειγμα, η δορυφορική, αν θέλετε, υποδομή που έχουμε σήμερα δεν μπορεί ε, να ανταποκριθεί ε, στις ταχύτητες που έχουμε σήμερα, αλλά μπορεί σε 10 χρόνια ναι. Έπειτα, τα κενά στον εφοδιασμό δείχνουν ότι ήδη είμαστε πολύ πίσω από τους ανταγωνιστές μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό λόγω των ε, εξελίξεων στο cloud computing. Το cloud computing απαιτεί μια πιο συμμετρική ανάπτυξη των ευρυζανικών υπηρεσιών. Γιατί λοιπόν αυτό είναι σημαντικό. Η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο την επόμενη 20 ετία, 30 ετία από το cloud computing. Και πάμε παρα... Πέρα, βλέπετε μια επανάληψη ουσιαστικά. Βλέπετε την Ιαπωνία και την Κορέα αριστερά στι στήλε. Είναι στοιχεία του ΟΣΑΜ και βλέπετε ότι τα πιο πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης υπολείπονται σημαντικά από τον μέσο όρο του ΟΣΑΜ. Βλέπετε τις χώρες της Βαλτικής που πηγαίνουν καλύτερα από τον μέσο όρο του ΟΣΑΟ. Π.χ. Σλοβακία επίσης βλέπετε. Γιατί προσαρμόστηκαν πολύ ε, γρηγορότερα αυτές οι χώρες, ιδίως ε, στην τεχνολογία των οπτικών ινών. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια και στους ε, τομεακούς στόχους. Για να έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος και του περιβάλλοντος, στην ενιαία αγορά, συν ε, την επίτευξη των στόχων ε, της ψηφιακή ατζέντα, ώστε το 2020 να έχουμε πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους έως τα 30 Mbps και πρόσβαση στο 50% των νοικοκυριών στα 100 Mbps. για να έχει μεγαλύτερη δυναμική αγορά ως προς το να επενδύσει σε, στις ευζωνικές υπηρεσίες. Και να είναι πιο εύκολη η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουν και τα κράτη-μέλη για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε διασυνδέσει ανάμεσα στις υφιστάμενες πλατφόρμες των κρατών μελών. Δηλαδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες πλατφόρμες που να αντικαταστήσουν τις εθνικές που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση. Δεν έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Επιχειρησιακή στόχη. Εδώ επαναλαμβάνω ουσιαστικά αυτά που ήδη είπα και νωρίτερα για την βιωσιμότητα των ε, ευρυζωνικών project. Και πρώτη, δεν, μάλλον, όταν δεν υπάρχει business case, πώς θα παρέμβουμε. Προχωρώ γρήγορα στην επόμενη διαφάνεια για τη λογική της πολιτικής μας, το συλλογισμό μας, σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές. Λοιπόν, πού θα παρέμβουμε. Αστικά κέντρα δεν είναι προτεραιότητα γιατί οι αγορές κατά πάσα πιθανότητα θα ρυθμίσουν τα των αστικών κέντρων τα επόμενα έτη. Μα ήδη έχει καλύψει τα πιο πολλά ε, κενά και ανάγκες. Αν πάτε σε πόλεις όπως η Στοκχόλμη, Ήδη έχετε το FTTH. Σε, στα προάστια, στα ημιαστιακά κέντρα, εξαρτάται από τον βαθμό ε, τη ε, κατά πόσο είναι πυροκατοικημένε, κατά πόσο υπάρχει διάθεση για επενδυσεις απο από κράτη-μέλη ή από άλλους φορείς που επενδύουν, όπως οι τηλεπικοινωνικές ε, εταιρείε, εταιρείε κοινή ωφελία, η ΟΤΑ κτλ. Στις αγροτικές περιοχές δεν υπάρχει αυτή Σήμερα στις αγροτικές περιοχές ε, γιατί μιλάμε. Για ε, 2.500 ευρώ αναγραμμή είναι το κόστος για να συνδεθεί ένα νοικοκυριό ε, και δεν θα καταβάλει αυτό το κόστος η αγορά. Δικαιούχοι του ΣΕΦ τηλεπικοινωνικέ εταιρείε, εταιρείε κοινής περιφερειακοί φορείς όπως και δήμοι και νέες συμμαχίε. νέες επενδυτικές εταιρείε που ε, συστήνονται ad hoc για να συμμετάσχουν σε προγράμματα του ΣΥΦ, εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα PPP δηλαδή. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια πού είναι τα αποτελέσματα μία ε, μελέτης που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και δίνει μία σειρά περιπτώσεων, σεναρίων που είναι πολύ πιο φιλόδοξα από αυτό που θέλουμε εμείς. Και σχέση με τα πιο φιλόδοξα σενάρια, μιλάμε 221 δις σε ανάγκη επενδύσεων. Αυτό τι θα σήμαινε, για παράδειγμα, να καλυφθούν περιοχές που ήδη καλύπτονται από τις αναλογικές υπηρεσίες. Βεβαίω αυτό είναι κάτι που απασχολεί κάποια κράτη-μέλη. Δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες, τις ενσύρματες όλα τα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Λογική πολιτική για τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών. και για, τον, για το στρώμα της πολιτικής που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το e-gov, ε, την ηλεκτρονική υγεία κτλ. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες επίσης. Υπάρχει και το PetPol που είναι ένα πιλωτικό project για αυτό το τομέα ήδη και υπολογίζουμε ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε περίπου 50 δις ευρώ επιτρέποντας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν προσβασιμότητα μέσω των τοπικών εμπορικών τους επιμελητηρίων και να έχουν διασύνδεση με άλλα αντίστοιχα επιμελητήρια ώστε να γίνονται τα γραφειοκρατικά στοιχεία πολύ πιο εύκολα όταν υπάρχει ιδιοσυνοριακό εμπόριο στις υπηρεσίες. Έξυπνα δίκτυα. Αυτό αφορά βεβαίως και την ενεργειακή συνιστόσα του ΣΕΦ. Για τις οπτικές ε, ίνες χρησιμοποίησαμε τους έξυπνους μετρητές και δημιουργήσαμε συνέργειες με το, την ενεργειακή συνιστόσα του Connecting Europe. Όπως η κυρία Γκάλο μας είπε ήδη, υπάρχουν και υπηρεσίες που δεν ε, δίνουν τόσο έμφαση στην οικονομική συνιστόσα, αλλά είναι πιο, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, σε άλλου είδους, αν θέλετε, σκοπούς, εστιάζουν. Οπότε ε, γίνεται δουλειά και προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλες υπηρεσίες, το e-government που είπα και πριν, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που μπορεί να βοηθήσει πολύ αυτό το είδους η επένδυση για την παροχή πιο πολλών πληροφοριών, έπειτα υπηρεσίε ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή identification. Δηλαδή είσαι ένα άλλο κρατό μέλο και μπορεί παρά τα αυτά να κάνεις δραστηριότητες μέσω του τσίπ που έχεις στην ε, ηλεκτρονική σου ταυτότητα. Βέβαια σε χώρες που δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες, δεν υπάρχουν καν ταυτότητες, μπορείς να το κάνεις αυτό μέσω της άδεια οδήγηση ή άλλων συσκευών πρόσβαση πληροφορίες στο δημόσιο τομέα και ε, πολυγλωσσικές υπηρεσίες. Θα συμπεριληφθούν τις υπηρεσίες σε όλες τις προαναφερθείς υπηρεσίες, δηλαδή μετάφραση σε όλες τις γλώσσες κτλ. Αυτό είναι και ο πυρήνας της όλης υπηρεσίας για να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες. Θα σας σταματήσω, λέει ο Πρόεδρος, εδώ. Καλύψατε τους βασικούς τομείς σχετικά με το πρόγραμμα επενδύσεως και νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα που θέλουν να δουν οι κυβερνήσεις και θα ήθελα να κανονίσουμε μία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε και η, πτυχή της ενιαίας αγοράς και την παροχή ενιαίων υπηρεσιών είναι επίσης σημαντικό θέμα και όπως είπατε ο ρόλος των των δικτύων είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που ήρθατε και Λυπάμαι ότι καθυστερήσαμε, αλλά θα επιτρέψουμε στην ομάδα υπό τον κύριο Γκάλερ να το παρακολουθήσει και θα μας στείλετε μια έκθεση μέχρι ε, τέλος Μαΐου. Έκτοτε θα ξανασυναντηθούμε μαζί με τους κοιόδους εισηγητές σας και όσον αφορά τη συζήτηση της εκθέσεώς σας 21-22 Ιουνίου, τροπολογίες μέχρι τις 29 Ιουνίου και ψηφοφορία τον Οκτώβριο για να έχουμε αρκετό χρόνο να το επεξεργαστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Γκάλερ και ευχαριστώ και όσους παρίσταντο. Θέλω λοιπόν να πω τώρα στα μέλη της Επιτροπής να είναι εδώ στις 3 η ώρα για την πολύ σημαντική ακρόαση σε αυτή την αίθουσα σχετικά με τις επαγγελματικές ικανότητες και τα διπλώματα. Ευχαριστώ όσους παρέστησαν το κοινό και ευχαριστώ που μπορέσαμε και προχωρήσαμε σήμερα.